Ladies and gentlemen, Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας ως ήθιστε μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Η διερμηνία υπάρχει για τις γλώσσες των ε, τακτικών μελών της Υποεπιτροπής αυτής Ασφάλειας και Άμυνας. Αρχίζουμε με το πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο δεύτερο σημείο. Έχουμε διάφορα πρακτικά να εγκρίνουμε. Συγγνώμη που σας τα έχουμε υποβάλει κάπως αργά, αλλά είναι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 21ης και 22ης Σεπτεμβρίου του 2015. Πρώτα απ' όλα. Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να σας τα στείλουμε νωρίτερα. Τα κοίταξα κι εγώ πολύ προσεκτικά, δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο. Υπήρχε ένα διοικητικό σφάλμα και γι' αυτό υπήρξε η καθυστέρηση αυτή. Ζητώ και πάλι συγγνώμη. Έχουμε και άλλα τρία πρακτικά. 25 Ιανουαρίου του 2016 4 Φεβρουαρίου και 17 και 18 Φεβρουαρίου. Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτής μπορείτε να κάνετε παρατηρήσεις, σχόλια. Εφόσον δεν υπάρχουν σχόλια και παρατηρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Και τώρα Συνεχίζουμε. Περνάει στα πολωνικά η πρόεδρος. Θα περάσουμε στα συγκεκριμένα σημεία ουσίας που έχουμε να εξετάσουμε σήμερα στην υποπιτροπή μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να σας παρουσιάσω εδώ τους ομιλητές μας. Θα παρουσιάσουν μελέτη που ζήτησε η υποπιτροπή μας να γίνει και είναι η πρώτη παρουσίαση που θα γίνει. Την έχετε, δεν πρόκειται βέβαια για το επίσημο το τελικό και γι' αυτό δεν θελήσαμε να το έχουμε μοιράσει προηγουμένως το έγγραφο αυτό. Συνεχίζει στα αγγλικά η πρόεδρος. Έχουμε δύο αξιότιμα μέλη, τον ε, μέτρο Φρεντερίκ Μαουρό ο οποίος είναι στον ε, Δικηγορικό Σύλλογο της Γαλλίας και τον Χαστομά, που είναι καθηγητής, στο, και στην ε, στρατιωτική σχολή, τη γερμανική του Μονάχου. Θα μας παρουσιάσουν τη μελέτη αυτή λοιπόν που αναφέρεται στο μέλλον της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της άμυνας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν θα τους δώσω το λόγο. Έχουμε πολλά θέματα και το πρωί και το απόγευμα, οπότε μην καθυστερούμε περισσότερο. Πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο κύριος ε, Μωρό και μετά ο κύριος Στομά. Λοιπόν, έχετε το λόγο κύριε Μωρό. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε κυρία Φωτίγκα. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μας που είμαστε εδώ και μπορούμε να σας παρουσιάσουμε την μελέτη μας που φέρει τον τίτλο «Το μέρον της Ευρωπαϊκής Έρευνας στον τομέα της άμυνας». Είμαι καθηγητής ε, μηχανικής στο Μόναχο. Θα περάσω αμέσως με την επόμενη διαφάνεια. Όταν ξεκινάει την ανάπτυξη, ξεκινάει με ε, διάφορες ε, τεχνολογίες. Ξεκινάμε από το επίπεδο ετοιμότητας της τεχνολογίας. Όταν ξεκινάμε από το 0 ξεκινάμε με το TRL1, ενώ αν προχωρήσουμε σε υψηλότερα επίπεδα μπορούμε να καταλήξουμε ε, στην ανάπτυξη μιας τεχνολογίας. Και βλέπετε εδώ ομαδοποιημένες τις κατηγορίες. Έχουμε την έρευνα και τεχνολογία, R&T, και έρευνα και ανάπτυξη R&D. Ε, θα σας εξηγήσω αυτές τις ε, δύο έννοιες στην επόμενη διαφάνεια και αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά αποτελέσματα της μελέτης ε, που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Όταν βλέπουμε τα νούμερα, βλέπουμε σημαντική μείωση στην έρευνα, στην άμυνα από το 2006 μέχρι το 2013 ως ανελεύθερη πτώση. Ε, στο R&D, έρευνα και ανάπτυξη, κατεβήκαμε κατά 29% ενώ στην έρευνα και τεχνολογία είχαμε μείωση της τάξης του 28%. Και επίσης, εάν δούμε τη, συλλογικά την έρευνα και τεχνολογία διαφόρων χωρών, ε, βλέπουμε μείωση 8%. Άλλο σημαντικό στοιχείο που θα δείτε εδώ είναι η υψηλή συγκέντρωση ε, της έρευνας σε τρεις χώρες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία. Εάν προσθέσουμε τα ποσά βλέπουμε ότι δαπανούν περίπου το 92% γύρω στο 90% του συνολικού ποσού ε, για την ε, έρευνα και ανάπτυξη και έρευνα και τεχνολογία. Βλέπουμε λοιπόν σημαντική συγκέντρωση σε αυτές τις τρεις χώρες. Προχωρώ στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε κάποιες ε, φωτογραφίες για να καταλάβετε το τεχνολογικό κενό που υπάρχει το τεχνολογικό χάσμα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, είχαν το 2002 το πρώτο μη επανδρομένο αεροσκάφος ενώ στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία αντίστοιχη βλέπετε την πρώτη πτήση το 2012 λέει ο το 2013 για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε στη στις Ηνωμένε Πολιτείες το 2002. Έχουμε λοιπόν ένα τεχνολογικό χάσμα 10 ή 11 ετών. Αυτό είναι τεράστιο χάσμα σε αυτού του είδους την τεχνολογία. Τι να κάνουμε λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Θέλουμε στην έκθεσή μας να δείξουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, τη δουλειά μας ε, όπως ε, προχωρούσαμε μέχρι τώρα. Εάν συνεχίσουμε να προχωράμε με αυτούς τους βραδείς ρυθμούς μέσα σε 10 χρόνια, ε, η βιομηχανία άμυνας ε, θα είναι μια περιθωριακή ε, βιομηχανία και θα χάσουμε όλες τις τεχνολογίες εχμής. Αυτό θα έχει οικονομικές συνέπειες διότι θα χάσουμε τη βιομηχανική βάση μας στον τομέα της άμυνας και από πολιτικής πλευράς αν ακούσετε τις συζητήσεις όλοι μιλάνε για στρατηγική αυτονομία. Εάν όμως δεν έχουμε τεχνολογίες εχμής, εάν δεν έχουμε τις κρίσιμες τεχνολογίες, αυτό θα είναι απλά λόγια κενά. Επίσης, συχνά λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια και είμαι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση που να παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Εάν όμως δεν έχουμε τη στρατιωτική ικανότητα ε, δεν θα έχουμε ελευθερία δράσης, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τίποτα στον κόσμο. Όλα αυτά είναι αρνητικά. Αλλά πρέπει να κάνουμε και θετικές δηλώσεις ε, που βλέπετε στο κάτω μέρος της διαφάνειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει αντιδράσει. Έχουμε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου του 2013 όπου αναφέρεται ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στον τομέα αυτόν, ενώ η ομάδα σας, ο κύριος Γκάλερ εδώ κάθεται, ξεκίνησε ένα πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε πρόγραμμα ερευνητικό για την άμυνα που χρηματοδοτείται από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική αυτή η χειρονομία. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία για μια προπαρασκευαστική δράση. τέλη Φεβρουαρίου θα προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες, σε λεπτομέρειες και φυσικά ο σημαντικός στόχος μας είναι να έχουμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας για την άμυνα που να ξεκινήσει το 2021 και να προχωρήσει μέχρι το 2028. Έχουμε λοιπόν θετικές δράσεις και στην επόμενη διαφάνεια θέτουμε το ερώτημα γιατί να τα κάνουμε αυτά, θα ε, υπάρχει προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση είναι ναι. Εάν εξετάσουμε εδώ τα διάφορα σημεία, διαπιστώνουμε ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανή να συγκεντρώσει την κρίσιμη μάζα όπως ε, είπαμε αρχικά, ουσιαστικά τρεις χώρες ε, δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν, αλλά χρειαζόμαστε κρίσιμη μάζα αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Επίσης έχουμε το πλεονέκτημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση με περισσότερη ασφάλεια και λιγότερες διακυμάνσεις διότι βλέπετε ότι πολλές χώρες όταν ε, λείπουν χρήματα ε, τα παίρνουν από τον προϋπολογισμό για την έρευνα αλλά ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η Ένωση μπορεί να ε, προσφέρει αποτελεσματική διακυβέρνηση διότι έχει πείρα σε τέτοιου τύπου προγράμματα. Επίσης εφόσον όλες οι ευρωπαϊκές χώρες συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται και την ευθύνη και ελπίζουμε ότι αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να μειώσουμε το χάσμα στην τεχνολογία που υπάρχει. Και η τελευταία μου παρατήρηση στη διαφάνεια αυτή είναι ότι η δράση αυτή της Ένωσης θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο οργανισμών έρευνας και τεχνολογίες, ώστε να συνεργάζονται στον τομέα της ε, έρευνας για την άμυνα όπως ε, συνέβη στον τομέα της ασφάλειας σε κάτι που ξεκίνησε ο κύριος Ήλερ και άλλοι. Δίνω το λόγο στον συνάδελφό μου Φρεντερίκ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές κυρίες και κύριοι. Αν συμφωνήσουμε με την αρχή που λέει ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας για την άμυνα αποτελεί μια προστιθέμενη αξία όπως μας κατέδειξε μόλις και ο φίλος Τόμας εδώ τότε, τρεις ερωτήσεις έρχονται στο μυαλό μου και αυτές ακριβώς θέσαμε και στους αυτούς μας. Η πρώτη είναι ποιο θα πρέπει να είναι το μέγεθος ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού ε, ερευνητικού προγράμματος άμυνας. Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος του και κατά πόσο ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να το συμπεριλάβουμε μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο δράση για την άμυνα. Α αρχίσουμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Ποιο θα πρέπει να είναι το μέγεθο ενό μελλοντικού ευρωπαϊκού προγράμματο έρευνα στον τομέα τη άμυνα. Θα είμαι ειλικρινή μαζί σα. Δεν υπάρχει τεχνική απάντηση σε αυτό. Κανένα εμπειρογνώμων δεν θα είναι σε θέση να σα απαντήσει. Η ερώτηση είναι πολιτική, εξού και η απάντηση που είναι επίση πολιτική. Δηλαδή, ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικά μιλώντας. Και εσείς είσαστε οι μόνοι που μπορούν να απαντήσουν αυτή την ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, θα σας δώσουμε και εμείς κάποια στοιχεία και περνάω στην επόμενη διαφάνειά μου. Όσον αφορά το συνολικό περιβάλλον, ας θυμηθούμε κάποια νούμερα. Υπάρχει η τρίτη πρωτοβουλία offset, βάσει της οποίας οι Ηνωμένε Πολιτείες αποφάσισαν να ξοδέψουν 64 δισεκατομμύρια το χρόνο τα επόμενα χρόνια για την έρευνα και την ανάπτυξη. Στην Κίνα κάπου 20 δισεκατομμύρια εκτιμάμε, πολύ συντηρητικά μιλώντας. Όσον αφορά τη Ρωσία, 3,54 δισεκατομμύρια για την έρευνα και την ανάπτυξη στην ε, άμυνα. Κάτι όμως που δείχνει ότι έχει διπλασιαστεί το ποσό τα τελευταία χρόνια. Αν συγκρίνουμε το 2013 στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές χώρες μόνο 7 δισεκατομμύρια έχουν δαπανηθεί για τον ίδιο σκοπό για την έρευνα και την ανάπτυξη δηλαδή και 2,1 δισεκατομμύρια για την έρευνα και την τεχνολογία. Όσον αφορά τώρα τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ε, τους διάσκεψης του ΝΑΤΟ του 2014 που ήταν 1,2 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο πρέπει να ξοδέψουν πολύ περισσότερα κάθε χρόνο και αν αυτό το αναλύσουμε όσον αφορά το R&D και R&D σημαίνει 1,2. Συνεπώς, πρέπει να γίνουν τεράστιες προσπάθειες από τις ευρωπαϊκές χώρες. 2,1 δισεκατομμύρια το χρόνο τώρα, συν 1,2 το χρόνο που έχουν αναλάβει την υποχρέωση να το κάνουν, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξοδεύουν 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι το ποσό που θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στην οικονομική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μείνει στο ίδιο επίπεδο, να μείνουν όλες οι χώρες στο ίδιο επίπεδο συνολικά. Το ελάχιστο επίπεδο τώρα για ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα άμυνας θα πρέπει να είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, που είναι αυτό που δαπανούν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνα στην ε, άμυνα, κάτω από το ποσό αυτό, δεν αξίζει το όνομα. Γιατί δεν μπορεί να αποφέρει καρπούς. Συνεπώς η επιλογή είναι ανάμεσα στα δύο αυτά ωραία, τα 3,3 δισεκατομμύρια και τα 500 εκατομμύρια. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε. Δεύτερη ερώτηση ποιο θα, ποιος θα πρέπει να είναι, ποιο θα πρέπει να είναι το αντικείμενο ενός τέτοιου ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνα στην άμυνα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο τεχνολογικός αγώνας είναι ένας αγώνας για να κερδίσουμε χρόνο, αν βρούμε στα πλαίσια του σημερινού πλαισίου, αυτό θα ήταν το πιο ρεαλιστικό. Συνεπώς, ως πρώτο βήμα για τα έτη για τα πρώτα έτη που πρέπει να τροποποιήσουμε, που θα ήταν το 2018-2020, υπολογίζουμε ότι υπάρχει διτή χρήση στην επιστήμη και την τεχνολογία μέσα στα πλαίσια του Horizon 2020 και ότι πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει ειδική στήριξη σε υποδομές και σε ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες ειδικού ενδιαφέροντος για την αμυντική κοινότητα. Αν δεν υπάρξει αλλαγή στον ορίζοντα 2020 στο νομικό του πλαίσιο, μπορούν να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Το επόμενο στάδιο που είναι το 2021-2028, εδώ πρέπει να υπάρχει ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας στην άμυνα που να βασίζεται σε τεχνολογικές μελέτες που να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να μειωθεί ο τεχνολογικός κίνδυνος για τις προμήθειες των χωρών μελών πρέπει να μειωθούν οι τεχνολογικοί κίνδυνοι. Και συγχρηματοδοτημένα προγράμματα επίσης θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με τις χώρες μέλη για να καλυφθεί το χάσμα ανάμεσα στα προγράμματα και την έρευνα στην άμυνα. Και η τρίτη μου ερώτηση είναι... Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Πώς να συμπεριλάβουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας στην Άμυνα με ένα πρόγραμμα δράσης για την άμυνα. Δύσκολη ερώτηση. Αλλά ας δούμε τα κύρια σημεία. Πρώτον, είναι βασικό να συνδέσουμε το πρόγραμμα το ερευνητικό στην άμυνα με τις ανάγκες ικανότητας. Και όλα αυτά, η έρευνα δηλαδή δεν μας έρχεται από το κοινό, από το κενό υπάρχει προηγουμένως κάποιος σχεδιασμός. Πριν από την έρευνα για την άμυνα υπάρχει ο σχεδιασμός της άμυνας. Γι' αυτό και χρειάζεται κάποια στρατηγική. Είχαμε 48 στρατηγικά έγγραφα να αναλύσουμε για να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας και να σας δώσουμε τα στοιχεία αυτά. Ποιες είναι οι ανάγκες ικανότητας λοιπόν που πρέπει να συγκεντρώσουμε για να ικανοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας. Πρέπει να δείτε λοιπόν την αναλογία και μόνο τότε φτάνουμε στο ζήτημα της έρευνας στην άμυνα. Γι' αυτό και λέμε ότι η έρευνα στην άμυνα έχει γνώμονα την ικανότητα. Η διαδικασία προμήθειας λοιπόν πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική όθηση, δηλαδή πρέπει να λάβει υπόψη να αναλύσει ποιες είναι οι υπάρχουσες τεχνολογίες σήμερα. Και αυτό είναι κάτι που αποκτά όλο και περισσότερη σημασία όταν σχεδιάζουμε την άμυνα. Γιατί υπάρχει νέα σχέση ανάμεσα στην μη στρατιωτική και στρατιωτική έρευνα. Πριν η μη στρατιωτική έρευνα δεν ήταν όπως ε, σήμερα που εμπλέκεται με τη στρατιωτική. Γι' αυτό το νήμα των τεχνολογικών αναγκών πρέπει να το φτιάξουμε βάσει των αναγκών ικανότητας. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Όμως το πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως έχει σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δεν μπορεί να αναλάβει ένα μεγάλο πρόγραμμα. Πράγματι είναι για δύο λόγους. Γιατί είναι δύσκολο να σκεφτούμε ότι ο οργανισμός αυτός θα μπορούσε να θέσει τους προσανατολισμούς και να επιλέξει τα καλύτερα προγράμματα προς το συμφέρον όλων των χωρών μελών και βάσει της ομοφωνίας που ισχύει σήμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο ικανοποιητικά. Έπειτα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας πρέπει να επανδρώνεται παρκώς, να προσλαμβάνει δηλαδή ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν πολύ μεγαλύτερα προγράμματα, άρα χρειάζονται περισσότερα κονδύλια και όλοι γνωρίζουμε ότι ο προπολογισμό του οργανισμού αυτού έχει μπλοκαριστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό που είναι και το κατεξοχήν εργαλείο που διαθέτει και αυτό συστήνουμε εμείς να χρησιμοποιεί, τότε θα πρέπει να αλλάξει η διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και του σημερινούς κανόνες να αλλάξει και το μέγεθος του λειτουργικού προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να το κάνει αυτό ή δεν μπορεί να κάνει αυτή την τροποποίηση, τότε πρέπει να σκεφτεί άλλες λύσεις, όπως για παράδειγμα ε, μια ad hoc ε, κοινή επιχείρηση ή μια γενική διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ειδικό επίτροπο για την έρευνα στην άμυνα. Τώρα, πώς θα συνδέσουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνα στην Άμυνα με τα προγράμματα εξοπλισμών. Αυτό μπορεί να γίνει με συγχρηματοδότηση κάποιων μεγάλων προγραμμάτων με τις χώρες μέλη. Να συγχωνευτεί, για παράδειγμα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας με τον Κοινό Οργανισμό Συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά στην αρχή αυτός ήταν ο σχεδισμός, αυτή ήταν η ιδέα. Και αν έχετε την περιέργεια μπορείτε να διαβάσετε τα πρακτικά της ε, συνθήκης, της σχετικής, για να δείτε χωρίς καμία δυσκολία ότι αρχικά το σχέδιο ήταν αυτή η συγχώνευση. Και τέλος, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει διπλούς πόρους, αυτό θα ήταν μια λύση. Τρίτο στοιχείο, το πρόγραμμα θα πρέπει να δεχθεί τη συμμετοχή των χωρών μελών. Και αυτό είναι ζωτική σημασία, γιατί αν το πρόγραμμα αυτό θέλουμε να κάνει την αλλαγή, τότε πρέπει να συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη και όλοι οι φορείς εμπλεκόμενοι. Και θα γίνει αυτό αν επενδύσουμε στους ε, τομείς μεγαλύτερης στατιακής σημασίας στις χώρες μέλη, για να έχουμε προγράμματα τρίτου επίπεδου. Έπειτα πρέπει να στηρίξουμε και τους πιο δύναμους κρίκους στον τομέα της έρευνας στην άμυνα, τους οργανισμούς τεχνολογικής έρευνας, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τις επιχειρήσεις και καινοτόμους παντός Τέταρτο σημείο. Το πρόγραμμα πρέπει να δώσει κίνητρα και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να παίξει το ρόλο της. Συνεπώς, πρέπει να πάψουν να υπάρχουν οι φόβοι στον κλάδο που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει όμως ότι χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις και ότι στις επενδύσεις αυτές θα ακολουθήσουν ε, πραγματικά και σωστά προγράμματα εξοπλισμού. Με άλλα λόγια, όταν κάνουν ε, έρευνα, όταν η βιομηχανία κάνει έρευνα, να μην την κάνει έτσι για να την κάνει, να ξέρει ότι θα έχει αποτελέσματα. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο αυτό συστηματικά και να δημιουργήσει και να ενισχύσει αυτόν τον ε, κρίκο που λείπει, να συνδέσει δηλαδή τη συνολική στρατηγική με, κάτι που είπε και η κυρία Μογκερίνη, με το νέο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων. Η Ευρώπη δηλαδή πρέπει να ετοιμάσει μια νέα υποστρατηγική άμυνα ή μια λευκή βίβλο, αν θέλετε, για να καθορίσει τα επίπεδα φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα. Εν κατακλείδη, μια δράση σημαντική και αμέσως χρειάζεται στον τομέα της έρευνας στην ε, άμυνα. Είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλουμε να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα στην στρατηγική αυτονομία. Από πλευράς του ΝΑΤΟ ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι πρόσδεκτο και είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσει που έχει η Ευρώπη απέναντι στην συμμαχία οι χώρες μέλη πρέπει να έχουν την ευκαιρία να διασφαλίσουν την ελευθερία και την ε, δράση τους με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Για ένα τέτοιο πρόγραμμα λοιπόν θα είναι μια πραγματική στιγμή ειλικρίνειας, αυτό που ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες πράγμα, που σημαίνει να κάνουμε τα λόγια μας πράξη. Και εδώ θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου αυτή παραθέτοντας ε, έναν Αμερικανό που συνέταξε μεταξύ άλλων το Σύνταγμά μας, τον Πάτρικ Χένρικ, που είπε ότι ενωμένοι στεκόμαστε όρθιοι, ενώ διχασμένοι πέφτουμε. Ας ε, μην κατακαιρματιστούμε δηλαδή, γιατί κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε την ε, ένωση από την οποία εξαρτάται η ίδια ύπαρξή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πειθαρχημένη παρουσίασή σας θα έχουμε και δευτερολογίες. Αρχίζουμε όμως πρώτα συζήτηση ο Καλά πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τωμά και κύριε Μαωρό για την παρουσίαση αυτή είμαι ευγνώμων που μας παρουσιάσατε σήμερα εδώ τη μελέτη σας. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Timely θα λέγαμε στα αγγλικά. Ταιριάζει απολύτως στο πολιτικό πλαίσιο το οποίο μας περιγράψατε. Τον Ιούνιο η κυρία Μογκερίνη θα μας παρουσιάσει τη στρατηγική σας ε, και μετά θα υπάρξει λευκή βίβλος για την άμυνα και επίσης ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης. Μας περιγράψατε και την πραγματικότητα που ζούμε αυτή τη στιγμή και μας προειδοποίησατε ότι εάν συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτόν σε δέκα χρόνια ε, η βιομηχανία άμυνας της Ευρώπης ε, θα είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν θα είναι πια σε θέση να καλύψει τις δικές μας ανάγκες. όταν κοιτάμε τα νούμερα άλλων εταίρων ή ανταγωνιστών οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν ε, την πρωτοβουλία, την τρίτη πρωτοβουλία offset. Είναι η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για διατήρηση της ε, τεχνολογικής της προόδου. Θέλει να συνεχίσει να είναι 10 χρόνια μπροστά από όλους τους άλλους με την πρωτοβουλία αυτή και πιστεύω ότι ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε που θέλουμε να πάμε. Μας αναφέρατε την προστιθέμενη αξία που μπορεί να υπάρξει από την ε, έρευνα, από την αμυντική έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται η κρίσιμη μάζα όπως είπατε, χρειάζεται η χρηματοδότηση για ένα πολυετές πρόγραμμα και θα πρέπει να φροντίσουμε να αποκτούμε περισσότερη αξία από τα χρήματα που δαπανούμε. Στις παρούσες εξελίξεις ε, στο παγκόσμιο σκηνικό δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κατάσταση, θα πρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα και το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να μας δείξει ποια θα είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε εθνικά συστήματα. Σε πολλά Υπουργεία Αμήνης ή Οικονομικών υπάρχουν πολλοί έξυπνοι άνθρωποι που θεωρούν ότι α, εντάξει, αν κάνουν κάτι οι Ευρωπαίοι μπορούμε εμείς να εξοικονομήσουμε τα αντίστοιχα χρήματα. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να διαπιστώσουμε ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία και να εργαστούμε με αυτόν τον προσανατολισμό. από το πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε πέρσι και φέτος θα πρέπει να προχωρήσουμε στην προπαρασκευαστική δράση και να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για την επόμενη τριετία. Θα πρέπει να δούμε κατά το επόμενο διάστημα, ε, κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, Ποια λύση θα επιλέξουμε. Η Κομισιόν θα θέλει να έχει γενική διεύθυνση για την αμυντική έρευνα ή θα θέλει στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2021-2028 να κάνει κάτι ή μήπως να έχει μια κοινή δράση αν θεωρηθεί ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Είμαι ανοιχτό σε λύσεις, ε, θα πρέπει όμως να μην χάσουμε από τα μάτια μα τον στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχω κάποιες σκέψεις να σας αναφέρω. Το 2003, όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά, ήμασταν αρκετά μετροεπαθείς στι ε, φιλοδοξίε μα και είχε μόνο μία ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. Τώρα που είμαστε σε καλύτερη κατάσταση και όλοι αυτοί το, το αναγνωρίζουν, θέλω μια παγκόσμια στρατηγική. Μήπως αυτό όμως δείχνει ότι προσπαθούμε να καλύψουμε σαν αδυναμίε μα με μεγαλοστομίες. Αυτό να μας απασχολήσει. Άλλο ένα στοιχείο να αναφέρω λέει η μελέτη σας ότι εντάξει θα πρέπει να προχωρήσουμε και ότι δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση. Εντάξει, το παραδέχομαι δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση. Και είναι καλό που λέτε ότι αυτός είναι ένας τομέας όπου πραγματικά υπολοιπόμεθα εμείς. Για να απαντήσω όμως στο ερώτημά σας για το μέλλον της ε, έρευνας αυτής για την άμυνα να πω ότι εξού σημαντικό είναι και το μέλλον των δαπανών σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Να περάσω τώρα σε αυτά τα κίνητρα που αναφέρατε. Η τεχνολογική αυτονομία επαρκεί ως κίνητρο για να αρχίσουμε να επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη της μη που την έχουμε παραμελήσει τόσα χρόνια. Τι να σας πω. Η τεχνολογική αυτονομία σημαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι θα θέλαμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ρωτάω λοιπόν, εμείς θέλουμε πραγματικά να δράσουμε. Πού είναι η πολιτική βούληση που θα μας οδηγήσει στο να δράσουμε και να δούμε δηλαδή κατά συνέπεια ότι μας λείπει η ικανότητα και μετά να επενδύσουμε σε αυτή την ικανότητα και να δράσουμε. Όλα αυτά λοιπόν τα ερωτήματα, εκτός από το τεχνικό κομμάτι του θέματος που αναφέρατε, θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Να σας πω επίσης ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή πολιτική άμυνας και κατά συνέπεια κοινή έρνα και ανάπτυξη για την άμυνα της Ευρώπης τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε πολλαπλές απειλές Πολλές απλές αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να συμμετάσχουν εδώ, να εμπλακούν, αν θέλετε να είμαστε επιτυχείς. Όλοι πρέπει να συμμετάσχουν. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάποιες χώρες στη Δύση δεν θέλουν να ανταποκριθούν και τόσο σε αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Ευρώπη, απειλές δηλαδή, τότε πώς να πούμε σε αυτές τις χώρες ότι ό,τι και να αποφασίσουμε θα πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι. Εσείς είπατε σωστά για κάτι άλλο, ότι αν αποφασίσουμε αύριο να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για την έρευνα και την ανάπτυξη στην άμυνα, τότε έχουμε ικανά εργαλεία και θεσμούς να μας συνοδεύσουν σε αυτή την προσπάθεια και να μας δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα παρελκόμενα ερωτήματα νομίζω στην μελέτη σας που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο. Σμπουχνέρ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημερωτική σας εισήγηση. Για τη χρηματοδότηση θα ρωτήσω εγώ όλου του προγράμματος. Εσείς αναφέρετε τον ορίζοντα 2000 κάτι όπου θα υπάρξουν κάποια χρήματα που θα μεταφερθούν από εκεί. Οπότε καταλάβα, έχουμε να κάνουμε ένα πολιτικό, μη στρατιωτικό δηλαδή πρόγραμμα. Τα λεφτά τότε από πού θα έρθουν. Αν μιλάμε για κάποια προγράμματα που θέλουμε, τώρα θα πρέπει να γνωρίζουμε από πού θα λάβουμε τα κονδύλια. Θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες πληροφορίε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Έλλερ. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς και εγώ και να πω και εγώ πως και ο κύριο ότι είναι τεράστια προσπάθεια που κάνατε. Αν δούμε το παρελθόν νομίζω θα μας βοηθήσει. Όταν ξεκινήσαμε συζητήσεις για τα προγράμματα άμυνας, πολιτικής άμυνας, τότε είχαν πραγματικά όρεξη για τέτοιες πολιτικές, ήμασταν φιλόδοξοι, τα κοιτάξαμε όλα αυτά, υπάρχει βούληση, υπάρχει ελεγγύη κλπ. κλπ. Στην πράξη, αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή ως εσωτερικές πολιτικές ε, ασφάλειας, συνεργασία, η Frontex, εποπτεία των λιμένων, όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν βασίζονται σε αυτά που κάνουμε στα πλαίσια του προγράμματος ασφάλειας, έρευνας ασφάλειας. Βέβαια προχωράμε αργά, όπως ξέρετε, ένα βήμα μπροστά δύο πίσω, αλλά αν αυτό δεν το είχαμε κάνει πριν από 10 χρόνια, τότε στην ουσία δεν θα είχαν ταπανηθεί καθόλου χρήματα για κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις. Θα είχαν χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, στα πλαίσια ενός πολιτικού πλαισίου. Κάπου περισσότερο, αλλού λιγότερο αλλά αν δεν υπήρξαν αυτά που κάναμε πριν από 10 χρόνια θα είχαμε τίποτα. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πρώτο δίδαγμα από το παρελθόν. Δεύτερον, έστω και αν δεν μιλάμε για την άμυνα, σε πρακτικούς όρου αυτό που θα συμβεί θα είναι το εξή. Δεν θα έχουμε πια καθόλου σουηδική αμυντική βιομηχανία, αυτό θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα, ούτε πολωνική ας πούμε, και μην υποτιμάτε το ότι Μπορεί να μην είχαν πλήρως ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία όπως η Σουηδία, αλλά είχαν μια σημαντική βιομηχανία γιατί συμμετείχαν σε προγράμματα όπως το Airbus, το Airbus ή και άλλα προγράμματα. Οπότε θεωρώ ότι εδώ είναι το βασικό ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει πολύ πέρα από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία που είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη από ό,τι νομίζουμε και όπως είπαμε στο παρελθόν Έχουμε τελείως διαφορετικό πλαίσιο τώρα με την αλληλοκάλυψη μη στρατιωτικής τεχνολογίας και αμυντικής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για την κατασκευαστική δυνατότητα όσον αφορά την άμυνα, τη βιομηχανική μας δυνατότητα όσον αφορά την άμυνα και τις βασικές τεχνολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας αγοράς. Από την σκοπιά λοιπόν της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας, τον οποία εκπροσωπώ ο συντονιστής, αν δεν θέλουμε λοιπόν να επενδύσουμε σε αυτό, τότε θα μείνουμε μάτια χέρια. Γιατί μπορεί να υπάρξει σύμπραξη βιομηχανιών στην Ευρώπη, κάτι το οποίο μπορεί να μας ε, χαροποιεί. Ήδη βλέπουμε ότι στην Γαλλία είχαμε κάποιες εξελίξεις στον τομέα της ε, αεροναυπηγικής. Τα έχουμε λοιπόν συγχώνευση βιομηχανιών οι οποίες θα υποχρεωθούν να το κάνουν αλλιώς δεν θα επιβιώσουν για τις προμήθειες. Σωστά αυτά που είπατε για την πολιτική βούληση κλπ. Σωστά. Αλλά αν τώρα δεν επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία τότε μπορεί να μην υπάρξουν καθόλου επιλογές για μας. Και τι κάνουμε τώρα. Να αγοράζουμε Ισραηλινή, Αμερικανική τεχνολογία για τα drones. Αλλά μας λένε οι Αμερικανοί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ότι θα πρέπει να συμβάλλει τεχνολογικά περισσότερο η Ευρώπη και η συμμετοχή των Αμερικανών πούμε, σε οπτικές ίνες ή σε άλλους τομείς η συμμετοχή τους είναι σε συνάρτηση με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Δεν μπορούμε να είμαστε λοιπόν σωστοί εταίροι στο ΝΑΤΟ αν δεν έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία και μηχανία. Στρατηγικά λοιπόν το ΝΑΤΟ είναι κάτι το λογικό αν θα πρέπει να υπάρχει συμβολή, όταν μάλλον υπάρχει συμβολή και των Ευρωπαίων και δεν βασίζεται αποκλειστικά στους Αμερικανούς. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε και να δούμε τι γίνεται με τις προμήθειες, με τις συγχωνεύσεις κλπ. Αλλά ξαναλέω, χωρίς επενδύσεις σε αυτό το τομέα, τότε αν δεν γίνουν επενδύσεις σε αυτό το τομέα, τότε θα χάσουμε τα πάντα. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Ντονζόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Τουμάκη ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι τρεις στην συνάδελφοι. Για το στρατηγικό θέμα, συμφωνώ με τον κύριο Πασκού, δηλαδή όταν μιλάμε για αυτή την ικανότητα της στρατηγικής της Ευρώπης, θα πρέπει καταρχάς να γνωρίζουμε για ποιο πρόγραμμα μιλάμε. Έτσι. Επειδή αν δεν καθορίσουμε, αν δεν χαράξουμε προγράμματα, οι βιομήχανοι δεν θα ακολουθήσουν. Και τι θα κάνουμε αυτά τα προγράμματα. Αυτό είναι το τελικό μεγάλο ερώτημα. Τι θα κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό. Και συμμερίζουμε την άποψη λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι μεγάλες οι μεγάλοι θεωρητικοί λιγμοί έχουν ξεκινήσει όσον αφορά την παγκοσμία στρατηγική. Ωραία, πολύ καλά όλα αυτά καλύτερο να έχουμε κάτι τέτοιο από το να έχουμε τίποτα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια στρατηγική με σωστά καθεσμένε προτεραιότητε που δεν ισχύει ακόμα και θα πρέπει να υλοποιηθεί. Αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά και νομίζω ότι η αντίληψη των κυβερνώντων σε κάποιες χώρες έχει αλλάξει. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν στο οποίο βρισκόμαστε όσον αφορά την και την, καινοτομία. Δεύτερο σημείο το οποίο είναι βασικό είναι το δημοσιονομικό. Εμείς είμαστε πεπισμένοι. Και μιλάτε λοιπόν σε κάποιους που είναι πεπισμένοι, αλλά θα πρέπει να πείσουμε εξίσου και τους αδέλφους στον προπολογισμό. Εδώ, στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια γραμμή στον προπολογισμό. Αυτό δεν είναι μόνο διαδικαστικό, είναι πολύ πολιτικό ζήτημα όταν βλέπουμε ότι κάποιες άλλες προτεραιότητες ανακύπτουν και είναι πολύ δύσκολο να αρπάξει κανείς ε, κάποιο εκατομμυριάκι ή κάποια εκατομμύρια από εδώ και από εκεί από θέματα όπως το προσφυγικό ή από τα παραδοσιακά ζητήματα της Ένωσης η Γεωργία ή τα διευθυντικά τομεία που παραμένουν ισχυρά. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια πολιτική μάχη για να επιβάλλουμε δημοσιονομικά κάτι το σημαντικό. Και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω. Τι θεωρούμε ως σημαντική δημοσιονομική συμβολή. Γιατί θα υπάρξει βεβαίως μια διάθεση να κάνουμε μια συμβολική κίνηση με κάποια εκατομμύρια που δεν θα επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν σωστά κάποια προγράμματα. Και δεν θα πρέπει να, αποτελεί βεβαίως, να αποτελούν κονδύλια που θα αντικαταστήσουν τις ε, δημοσιομικές προσπάθειες της μηχανίας και των χωρών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ένας μηχανισμός χρηματοδότησης ευρωπαϊκός θα περιπλέξει το έργο των βιομηχάνων. Αν λοιπόν έχουμε μια σημαντική αλλά συμβολική ένα συμβολικό αλλά σημαντικό ποσό ανάλογα με το πρόγραμμα το οποίο όμως θα περιπλέξει την αρχή του προγράμματος θα περιπλέξει τους ελέγχους πριν και μετά ή κατά διάρκεια των προγραμμάτων ξέρετε αυτά είναι δυσκίνητα επειδή ακριβώς ε, από τις Βρυξέλλες τότε θα έχουμε κάτι αντιπαραγωγικό θα μπούμε λοιπόν σε αυτή τη φάση όπου θα πρέπει να προσδιορίσουμε σωστά τι γραμμέ πάνω στι οποίε θα βασιστούμε. Και ο Χριστιαν, ο οποίο έχει σημαντική εμπειρία, αναφέρθηκε προηγουμένω στα προγράμματα ασφάλεια, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό προηγούμενο για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουμε εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει επίση να καθορίσουμε πολύ ακριβώ τα προγράμματα για τα οποία θέλουμε να διαθέσουμε κονδύλια και τι κονδύλια θέλουμε να διαθέσουμε γιατί εδώ ακριβώ έχουμε να κάνουμε την αποτελεσματικότητα όλου αυτού του εγχειρήματος. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κλείνουμε τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τους δύο εισηγητές να θα θέλουν να απαντήσουν στις σκέψη και ερωτήσεις που ακούστηκαν. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα πολύ να απαντήσω κύριε Πασκού στην παρατήρησή σας ε, γιατί ε, μια συνολική στρατηγική δεν είναι υπερβολικό, το χρειαζόμαστε πράγματι. Πιστεύω πως ναι, σίγουρα χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Ακούσαμε αυτό που είπε και ο κύριος ε, Ήλερ. Ο... Υπάρχει παγκοσμιοποίηση και εάν κοιτάξουμε απομονωμένα τον τομέα αυτόν, αυτό θα είναι σημαντικό λάθος μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο ανταγωνισμός είναι επίσης παγκόσμιος. Ε, κοιτάξτε τι γίνεται στον ε, τομέα των αυτοκινητοβιομηχανιών ε, από τις οποίες ζει η Ευρώπη. Κοιτάξτε τι κάνουν οι αμερικανικές εταιρείες. Ή σκεφτείτε τι θα γίνει αν η Google διεισδύσει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, έχουμε παγκοσμιοποίηση. Ε, αν δεν το προσέξουμε αυτό, σε πέντε χρόνια θα έχουμε χάσει την ευημερία μας. Γι' αυτό λοιπόν στο ορίζον 2020 και στο σύνολο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης ώστε ό,τι έχουμε χάσει να το ξαναοικοδομήσουμε. Στον τομέα λοιπόν ε, της αμήνης μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κύριος Σίλερ. Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη και δεν ε, αγωνιζόμαστε μόνο σε αυτόν τον τομέα. Ε, αγωνιζόμαστε γενικά για την επιβίωση της βιομηχανίας μας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν σαφώς παγκόσμιο το πρόβλημα και η, σχετική βιομηχανία, η συγκεκριμένη βιομηχανία αποτελεί σημαντικό μέρος του προβλήματος. Ε, αγωνιζόμαστε για την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Ίσως ε, θα μπορούσαμε στην έκθεσή μας να κοιτάξουμε ε, όχι μόνο ε, τις συγκεκριμένες τιμές αλλά μάλλον θα είχαμε ξεπεράσει τα όρια της μελέτης μας. Μετά είχαμε την ερώτηση σχετικά με τα κίνητρα και την τεχνολογική αυτονομία. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Πασκού σχετικά με την ε, στρατηγική αυτονομία. Η στρατηγική αυτονομία δεν είναι μία κενή έννοια. Ε, συνδυάζει τρεις ελευθερίες. Την ελευθερία δράσης, ε, την ελευθερία ε, αντίδρασης, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να παράγουμε, να διατηρήσουμε, να υποστηρίξουμε και να πολλούμε τα δικά μας όπλα. Εάν δεν είναι κανείς ε, ικανός να παράγει τα δικά του όπλα, ε, εξαρτάται από άλλους για το θέμα της δικής του άμυνας. Και πίσω από τις ελευθερίες αυτές ε, υπάρχει κάτι παραπάνω. Η Ευρώπη οικοδομείται σε τρεις σημαντικές αξίες. Η μία είναι η η ειρήνη, η ελευθερία, όλες οι ελευθερίες, και αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες ελευθερίες, και η τρίτη βασική αξία είναι η ευημερία. Η βιομηχανία αποτελεί μέρος του ονείρου αυτού. Εάν λοιπόν θέλουμε να διατηρήσουμε την στρατηγική αυτονομία μας, θα πρέπει να μπορούμε να παράγουμε τα δικά μας όπλα. Είδατε ε, την φωτογραφία των ε, συστήματων ΕΦΚΑΣ. Είδατε το αμερικανικό αεροσκάφος και τα βρετανικά και ε, γαλλικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αυτό ξεκίνησε πριν 15 χρόνια. Η επόμενη γενιά Εάν συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτόν δεν ε, θα μπορεί να παράγει αυτό το όπλο. Ε, κύριε, ήμουν υπουργός, οικονομ... Ε, αμήνης και τα γνωρίζω όλα αυτά. Αλλά εγώ θα... Οι ομιλητέ μιλούν παράλληλα. Συγγνώμη, χάσαμε την μισή πανέβαση. Ε, Εσεί είσαστε οι μόνοι που μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό ή είναι πολιτικό, απαντά κύριο Στομά. Ο, κύριος Μωρό, ο κύριος Τωμά. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να σκεφτούμε την ε, χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από τον ε, κατακαιρματισμένο τρόπο σκέψης. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με την κυβερνοασφάλεια, με τις κρίσιμες τεχνολογίες που είναι τεχνολογίες πολλαπλών σκοπών. Πάντως ε, είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και όσον αφορά την χρηματοδότηση. Νομίζω όμως ότι γενικά σε πολλά μέτωπα θα πρέπει να σκεφτούμε καινοτόμα. Για παράδειγμα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια ή τις κρίσιμες τεχνολογίες. Σκεφτείτε για παράδειγμα την βιομηχανία 4.0. Είναι κάτι που έχουμε αναπτύξει στη Γερμανία. Ε, ναι, οι Αμερικανοί ήδη βρίσκονται εκεί, αλλά ε, εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα να τους ανταγωνιστούμε. Και αυτό θα έχει μεγάλη σημασία και στη βιομηχανία άμυνας. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Ντονζό. Να απαντήσω στον κύριο Ντονζό στα γαλλικά. Αναφέρατε τρία ερωτήματα. Κέρια. Το πρώτο. Για τη στρατηγική δυνατότητα και τα προγράμματα. Να επανέλθω σε διαφάνεια για τη στρατηγική μετάβαση. Πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα στο στρατηγικό τομέα όπως κάνουμε έρευνα στο πολιτικό τομέα. Η έρευνα για την άμυνα δεν είναι άσκοπη. Όχι αυτή, την προηγούμενη, την προηγούμενη. Αυτή, αυτή διαφανή θέλω. Ναι. Εδώ και 50 χρόνια όλες οι μεγάλες χώρες και πιστέψτε με, εξετάσαμε όλα τα στρατηγικά, στρατηγικά έγγραφα στο παράρτημα της έκθεσης. Εξετάσαμε 48 στρατηγικά έγγραφα. ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Δανία, ΝΑΤΟ. Δεν κάναμε στην τύχη λοιπόν κάποια πράγματα. Πρέπει να καθορίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Έτσι, αυτό που λέμε global strategy. Ποιε είναι οι φιλοδοξίε μα. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε λοιπόν τις φιλοδοξίες με τα μέσα που πρέπει να συνάδουν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε μια λευκή βίβλο η οποία θα καθορίζει το επίπεδο βλέψεων στρατιωτικών. Δηλαδή, τι θέλετε να πετύχετε στρατιωτικά, τι μπορεί να κάνει η Ένωση στρατιωτικά. Στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη, στο 5, πολιτική ασφάλειας και άμυνα σκηνέ καθορίζουν κάποιες, κάποιους στόχους. Ποια είναι τα στρατηγικά μέσα λοιπόν εδώ. Συγκεκριμένη ερώτηση που χρειαζόμαστε λοιπόν για να πετύχουμε αυτές τις αποστολέ μας. Αυτή λοιπόν διάρθρωση μεταξύ παγκόσμια στρατηγική λευκή βίβλου, δυνατότητα ανάπτυξη ικανότητα και σα παρακαλώ διακόπτει ο μιλητή, μπορούμε να πάμε στην τελευταία διαφάνεια. Στο τέλος δηλαδή της παρουσίασης. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην τρέχετε τόσο γρήγορα. Πριν, πριν. Άλλη μια στο παιδό. Εδώ λοιπόν βλέπετε πώς διαρθρώνονται οι διάφορες φάσεις μιας στρατηγικής λογικής σε ένα σχεδιασμό άμυνας. Αν δεν έχουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία σε αλληλουχία και τα οποία θα μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται, τότε δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Αυτό λοιπόν αφορά και το άλλο ζήτημα για τους φίλους μας του, στα δημοσιονομικά που πρέπει να τους πείσουμε. Αλλά εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό ως κοινοβούλιο, να ψηφίσετε σε έσοδα. Εσείς είστε εκλεγμένοι από το λαό ερετή για να το κάνετε αυτό. Βέβαια θα είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν οι μορφές έτσι Μεσολάβηση που τέλο πάντων σας επιβάλλουν κάποιες επιλογές, αλλά μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. Τώρα, τι αποτελεί σημαντικό ποσό. Προσπάθησαμε να καθορίσουμε κάποια όρια όσον αφορά αυτές τις παρεμβάσεις και είπαμε ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από τι χώρε μέλη, τότε χρειάζονται δύο δις. Λίγο σε σχέση με τα 67 των Αμερικανών. Ελάχιστα. Λαμβάνοντα υπόψη ένα θετικό σενάριο όπου τηρώνται τέλος πάντων οι δεσμεύσεις διασκέψεων κορυφής στην Ουαλία και τα λοιπά το 14. Έχουμε λοιπόν καθορίσει το τι εκπροσωπεί για την κάθε χώρα η δέσμευση της Ουαλίας. Ένα δις. Ξέρουμε λοιπόν ότι η Ένωση δεν μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να αντικαταστήσει τις χώρες μέλη. Ποιο είναι το βασικό φάσμα, βασική δέσμη εδώ. Είναι αυτή λοιπόν που μας παρέχει η μεγάλη, μια χώρα όπως η Μεγάλη Βρετανία, 500 εκατομμύρια ετησίως, 540 Γερμανία, 550 ε, εκατομμύρια ετησίως η Γαλλία και αυτά είναι αυτά που θα πρέπει να δαπανηθούν ετησίως για να έχουμε ένα φάσμα σχετικά πλήρες. Νομίζω ότι δώσαμε μια σαφή απάντηση λοιπόν σε αυτό το ερώτημα της χρηματοδότησης. Κάτω από τα 500 δεν άξιζε τον κόπο. Γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο θα περιπλέξετε τις μηχανικές διαδικασίες και θα δημιουργήσετε έτσι κάποιες ασάφειες και θα πιστέψουν οι πολίτες ότι η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα και είναι καλύτερο να μην κάνει τίποτα από το να κάνει κάτι λίγο. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτά τα ποσά για να βοηθήσουμε τις ε, χώρες μέλη. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σέρλε ήθελε το λόγο για δευτερολογία. Παρακαλώ. Συγγνώμη που θα το πω έτσι στα ράτα. Αλλά όταν ξεκινήσαμε την, το πρόγραμμα για την ασφάλεια είμαστε στην ίδια κατάσταση. Μεγάλα προβλήματα με το Συμβούλιο, με την Κομισιόν, επειδή ήταν προετοιμασμένη, το Κοινοβούλιο το οποίο έχει αγανακτήσει. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια έκκληση εδώ στην αυτοπεποίθησή μας. Πρέπει να μιλήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο με όλες τις ομάδες, πολιτικές, για να δούμε τι γίνεται με τις προοπτικές. Αφιβάλλω να θα χρησιμοποιήσουμε έρευνα πούμε, για ένα ευρωπαϊκό τάγκ. Έχουμε καταστάσεις ασφάλειας που απαιτούν παρακολούθηση, υποπτία, συνδυασμό ασφάλειας και στρατηγικού χαρακτήρα. Έχουμε αποστολές, έχουμε αποστολές που θα πρέπει να προστατευτούν. Οπότε αυτή η διαλειτουργικότητα της Ένωσης έχει σχέση εδώ. Οπότε υπάρχει ένα κοινό πεδίο. Και μου είπαν κάποιοι άλλοι, κοιτάξτε, δεν θα πάρετε χρήματα για αυτό. Και συνέβη το αντίθετο. Τα πήραμε. Εντάξει, θα αλλάξουμε τον κόσμο. Νομίζω όμως ότι για, το επόμενο, για τα επόμενα χρόνια έχουμε 85 δις το 2% είναι 3 δις. Τόσο μακριά είναι αυτό από αυτό που διαπραγματευόμαστε με το Συμβουλίο. Δεν πιστεύω. Μπορούμε να το πετύχουμε λοιπόν. Υπάρχει τώρα το θέμα βέβαια το πολιτικό, αν υπάρχει πλειοψηφία γι' αυτό. Αν όμως θέλουμε πραγματικά μπορούμε να το πετύχουμε ως ποσό. Και νομίζω το Συμβούλιο έχει κατονόησει ότι κάτι πρέπει να κάνει η Κομισιόν επίσης, και πρέπει να τη βοηθήσουμε, και το Κοινοβούλιο είναι αλήθεια ότι είναι σε κάποια απόγνωση. Έχουμε έτσι την ε, νεμοποίηση του θύματος, έχουμε δίκιο αλλά χάνουμε. Λοιπόν, αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό δεν θα πάμε πουθενά. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να χαράξουμε αυτό το πρόγραμμα και να δώσουμε τα κονδύλια. και να πάμε στο Συμβούλιο και να αναζητήσουμε ένα συμβιβασμό. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ γιατί βρισκόμαστε αν δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη αν δεν συνεργαστούμε με άλλους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Με αυτά ασχολείται ή πρέπει να ασχολείται το Κοινοβούλιο Πονοπολογισμό, έρευνα, δικέ μα αρμοδιότητε. Και θεωρώ ότι αν υπάρχει ομόνια εδώ στην πλειοψηφία στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο, το θα μπορέσουμε να κάνουμε μια παρασκευαστική δράση και να χαράξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι εφικτό χωρίς να υποκαταστήσουμε εθνικές δράσεις ή να αντιγράψουμε τους Αμερικανούς, αλλά να κάνουμε κάτι ουσιώδες. Το έχουμε κάνει και μπορούμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πασκού. Θέλετε να απαντήσετε. Όχι. Εμένα η θέση μου ήταν ότι ακόμα και αν τα καταφέρουμε όλα αυτά, το πρόβλημα παραμένει. Και όπως προτείνατε, δεν τίθεται θέμα ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε. Μπορούμε ε, να ασχοληθούμε με την πολιτική πτυχή ε, και έτσι να φτάσουμε στην ε, στρατιωτική. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταφέρουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Και συμφωνώ μαζί σας ότι με το που ε, θα χάσουμε τις τεχνολογίες αυτές, ε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, ε, να τις ανακτήσουμε, να επιστρέψουμε στο σκηνικό. Ε, κυρίες και κύριοι, α, παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα... Να αναφέρω ότι η συζήτηση αυτή ε, ακούγεται μάλλον θλιβερή. Δεν είναι η πρώτη συζήτηση που έχουμε εδώ για το θέμα αυτό και δείχνει σαφώς ότι όταν μιλάμε για άμυνα και νέες τεχνολογίες ε, είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα ήθελα όμως να το δούμε υπό διαφορετική οπτική, διότι το πρόβλημα που βλέπουμε στην Ευρώπη γενικά, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο ότι δαπανούμε πολύ λίγα χρήματα στις νέες τεχνολογίες. Έχετε τα νούμερα τα οποία είναι ακριβή. Δυστυχώς όμως, οι πόροι αυτοί δεν δαπανούνται αποτελεσματικά. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Θα μπορούσαμε να θέσουμε την εξής ερώτηση. Δαπανούμε δισεκατομμύρια ευρώ και τι καταφέραμε με αυτά. Τι προγράμματα έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν λάβουμε υπόψη τις δαπάνες όλες αυτές. Μπορούμε να μιλάμε στο και για μία επιτυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εγώ θα πρότεινα την εξή λύση, διότι δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πείσουμε ο ένας τον άλλον. Χρειάζεται να είναι απαραίτητο να αυξήσουμε τους πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι από δύο δρόμους μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Καταρχάς, περισσότερους πόρους στην πολιτική έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από την προσέγγιση που βλέπουμε σήμερα που λέει ότι τα ποσά αυτά δεν μπορούν να δαπανηθούν ε, σε έρευνες ε, που να σχετίζονται με αμυντικές εφαρμογές. Νομίζω ότι αυτό είναι τελείως παράδοξο, διότι σε πολλές περιπτώσεις ε, μιλάμε για τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολιτικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς, για, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές εφαρμογές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την αρχή αυτή στα μελλοντικά προγράμματα και δεύτερον, θα πρέπει να εξετάσουμε τους πόρους και το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Ε, δυστυχώς δεν νομίζω ότι είναι πολύ αποτελεσματικός οργανισμός αυτός. Λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια. Έχει λάβει σημαντικά ποσά από τα κράτη-μέλη. Και μήπως θα πρέπει να θέσουμε ένα πολύ βασικό ερώτημα. Τι έχουμε πετύχει με όλα αυτά. Η απάντηση δυστυχώς είναι όχι πολλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας. Παρακαλώ. Ο κύριος Στομά, σας ευχαριστώ πολύ. Σημειώνω αυτά που είπατε. Μιλήσατε για τον αυστηρό διαχωρισμό που γίνεται ανάμεσα στην αμυντική και την άλλη έρευνα. Νομίζω ότι αυτό θα λυθεί. Αρκετοί μιλούν για έρευνες πολλαπλού σκοπού, όχι δηλαδή καθαρά αμυντική ή καθαρά βασική πολιτική έρευνα. Ιδιαίτερα για τα χαμηλά επίπεδα TRL δεν μπορεί να γίνει αυστηρά αυτή η διάκριση. Μιλάμε για βασικές τεχνολογίες στις περιπτώσεις αυτές, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς παντού. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε και ε, τα αισθήματα μας στο θέμα αυτό. Αν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τον αυστηρό αυτό διαχωρισμό, νομίζω ότι θα κερδίσουμε πολλά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Όταν βλέπουμε τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε σύντομα, Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι ειδικά στα χαμηλά επίπεδα TRL δεν θα πρέπει να γίνεται αυτή η αυστηρή διάκριση στα υψηλότερα επίπεδα τεχνολογίας ε, μπορεί να ε, πρέπει να γίνει η διάκριση, αλλά κάποιες τεχνολογίες ε, σίγουρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς λόγους. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα αυτό πράγματι. Κύριε, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα είναι ότι καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση, διότι έχουν εξαντληθεί τα χρονικά μας περιθώρια. Λυπάμαι πολύ. Σίγουρα θα επανέλθουμε στη συζήτηση αυτή, διότι φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευρά των βουλευτών. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν χαρά μας ε, που μιλήσατε εδώ στην ε, Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. I'm going first. Ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ. Παρακαλώ τους ευρωβουλευτές που δεν θέλουν να παραμείνουν στην αίθουσα για το επόμενο σημείο οι εμπειρογνώμονες αν θέλουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν σύντομα παρακαλώ. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ο τρίτος προσκεκλημένος έχασε το τρένο του από ό,τι φαίνεται και θα καθυστερήσει. Προσπαθούμε λοιπόν να οργανώσουμε εκ νέου τη σειρά των παρουσιάσεων. Το θέμα λοιπόν αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται για την προστασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών από την πειρατεία. Έχω λοιπόν το προνόμιο και τη χαρά εδώ να υποδεχτώ δύο διακεκριμένους προσκεκλημένους που γνωρίζετε πολύ από εσά. Ο πρώτος είναι ο κύριος Σάιμον Church, ο οποίος είναι αξιωματικός σύνδεσμος του κλάδου στο ΝΑΦΟΡ στη Σομαλία. Ο δεύτερος είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση ΜΟΦ που ειδικεύεται σε θέματα ναυτιλιακής ασφάλειας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Όταν φτάσει και ο κύριος Νόουξ, τότε θα κάνει και εκείνο τη δικιά του παρουσίαση. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα. Λοιπόν, κύριε Τσέρτς, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Ονομάζομαι Simon Church, είμαι αξιωματικό σύνδεσμος του κλάδου στο Νάφορ, στην Σομαλία. Δουλεύω βέβαια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις Νάφορ που είναι η Αταλάντα. Υπάρχει όντως διαφορά ανάμεσα σε μια στρατιωτική και μη στρατιωτική δράση αλλά υπάρχει σχέση ανάμεσα στο στρατιωτικό σκέλος και την ναυτιλιακό κλάδο. Στα 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου θα σας παρουσιάσω κάπως σύντομα που βρίσκεται το κέντρο ναυτιλιακής ασφάλειας όπου είναι το επιχειρησιακό κέντρο της ΝΑΦΟΡ, πώς λειτουργεί, πώς βοηθάει τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και μετά θα κάνω τη σύνδεση ανάμεσα τη δικιά μας δράση και την ναυτιλία. Η ναυτιλία φυσικά είναι το σημαντικό για μας, γιατί ακριβώ αυτό πρέπει να προστατεύουμε. Τα πλοία, τα σκάφη που κυκλοφορούν στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Πού βρίσκεται λοιπόν το κέντρο αυτό στο κέρας της Αφρικής. Θα δούμε και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να επικοινωνούμε, να μεταφέρουμε πληροφορίες. Θα σας εξηγήσω επίσης πώς στηρίζουμε και τη γενικότερη δράση κατά της πειρατείας. Όπως ίσως γνωρίζετε μερικοί από εσά, η, η UNAFOR είναι μόνο μία επιχείρηση από τις διάφορες που ισχύουν στον Δικό Κιανό σήμερα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και είναι ζωτική σημασία η επιχείρηση αυτή για την επιτυχία της όλης δράσης. Θέλω να επενθυμίσω σε αυτούς που δεν το γνωρίζετε ότι η εντολή για την επιχείρηση Αταλάντα άρχισε από το 2008 και βασίζεται σε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών του Συμβουλίου Ασφαλείας δηλαδή του ΟΙΕ. Το βλέπετε εδώ με κόκκινο ένας βασικός πυλώνας της αποστολής μας είναι η προστασία της ευάλωτης ναυτιλίας. Από την αρχή λοιπόν της αποστολής μας φροντίσαμε η σχέση μας με την ναυτιλία να αποτελεί και την προτερότητά μας. Ακριβώς επειδή ήταν προτερότητά μας καταφέραμε και να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη με τον ναυτιλιακό χώρο συνολικά, όπως θα δείτε και στη συνέχεια όταν σας παρουσιάσω τα μεγέθη, πόσα πλοία, πόσες επιχειρήσεις, πόσο προσωπικό χρησιμοποιούμε. Αυτή λοιπόν η βασική εμπιστοσύνη βοήθησε να αντιμετωπίσουμε την κρίση το 2009 όταν είχαμε 50 σκάφη που είχαν απαχθεί από πειρατές. 50 σκάφη το 2010 ένα τη βδομάδα περίπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εμπειρία συγκεντρώσαμε από την επιχείρηση αυτή. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε πετύχει στη συνέχεια, γιατί κερδίσαμε από αυτή την εμπειρία, βασιστήκαμε σε αυτή την εμπειρία και σχεδιάσαμε την συνέχεια της αποστολής μας. Λοιπόν, πώς ε, λειτουργεί αυτό το κέντρο ασφάλειας και προστασίας θαλασσίων εμπορικών οδών. Έχουμε το στρατηγείο μας, πρόκειται για μια στρατιωτική επιχείρηση και έτσι έχει οργανωθεί. Εμείς ανήκουμε στο επιχειρησιακό κέντρο, το GOC που είναι εδώ στον ε, κύκλο, που είναι το κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Σας είπα ότι πρόκειται για ένα κέντρο στρατιωτικό και μη στρατιωτικό έχει και τα δύο σκέλη συγχρόνως μαζί. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Είναι αυτή η μίξη των δύο διαστάσεων, της στρατιωτικής και τη μη στρατιωτικής. Εδώ λοιπόν βλέπετε ακριβώς το κοινό επιχειρησιακό κέντρο όπου απασχολούμαι και εγώ. Εδώ δουλεύω. Εφτά χρόνια και τρεις μήνες έχει που λειτουργεί δεν είναι ένα κλασικό κέντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι όμως ένα κέντρο που έχει και μη στρατιωτικούς οι οποίοι συνεργάζονται με αξιωματούχους της ναυτιλίας. Και η σχέση αυτή μας έχει επιτρέψει να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη από τον ναυτιλιακό χώρο. Αρχίσαμε να λειτουργούμε το 2009. Έχουμε 11.000 περίπου επιχειρήσεις οι οποίες είναι καταγραμμένες στο Ναυτιλιακό Κέντρο Ασφάλειας στο κέρος της Αφρικής. 4.500 σκάφη κάθε μήνα καταγράφονται γιατί περνάνε transit από την περιοχή. Συντονίζουμε λοιπόν και επικοινωνούμε με προειδοποίησεις προς τα σκάφη που βρίσκονται εν πλώ και έχουμε ένα μέσο τέτοιο προειδοποίησης. Τα σκάφη φροντίζουμε να μπορούν ασφαλώς να μετακινούνται. Συνοδεύουμε μερικές φορές τα σκάφη και είναι και ανεξάρτητοι οι οποίοι συνοδεύουν τα σκάφη αυτά που δεν αποτελούν μέρος του δικού μας κέντρου η Ιαπωνία, η Ινδία, η Κορέα, η Κίνα συνοδεύουν τα δικά τους, τις δικές αποστολές, τις ναυτικές, τα κομβόης πολλές φορές. Οι ίδιοι. Μέσω του μηχανισμού SAID επίσης γίνεται αυτό. Στον Μπαχρέιν κάθε τρεις μήνες έχουμε κάτι και θα έρθω σε αυτό αργότερα. Για να πάμε λίγο πίσω, παρακαλώ, στις διαφάνειες. Το πιο σημαντικό στοιχείο του κέντρου μας είναι ότι δημιουργήθηκε στα πλαίσια μιας κρίσης. Το ξεχνούν πολλές φορές οι άνθρωποι, αλλά η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη τότε. Και γι' αυτό και η UNFOR φρόντισε να συνεργαστεί και να ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη. Υπήρχαν εμπιστευτικέ πληροφορίες που είχαν τεράστια σημασία προκειμένου να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση και να προστατεύσουμε τα εμπορικά σκάφη. Συγχρόνως, όμως, έπρεπε να διασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν ασφαλείς, παρέμεναν απόρριτες. Συνεπώς γίνονται μεγάλοι έλεγχοι για να μπορούμε να διασφαλίσουμε την αυταλία ότι οι πληροφορίες τους είναι ασφαλείς μαζί μας. Και έτσι οικοδομήθηκε η εμπιστοσύνη στην οποία αναφέρθηκα πριν και βρίσκω τόσο σημαντική. Τι βλέπετε εδώ τώρα. Εδώ βλέπετε το σύστημα επικοινωνίας Mercury είναι ένα μη, για μη διαβαθμισμένες πληροφορίες που επιτρέπει επικοινωνία ε, σε πραγματικό χρόνο. Το έχουμε το σύστημα από το 2009 και το χρησιμοποιούμε έκτοτε συνέχεια. Χωρίς αυτό, άλλες δράσεις στον δικό κενό δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Έχουμε όλο και περισσότερα μέλη συμμετέχουν και οι αρχές συμμόρφωσης και επιβολής του νόμου των χωρών μελών, για παράδειγμα, πέρα από τους ε, ομολόγους μας. Συμμετέχει η Κένια, η Ινδία, το Αμάν και πολλοί άλλοι. Είναι πολύ βασικό το σύστημα αυτό και από πλευράς τακτικής και στρατηγικής για να ε, πετύχουμε στις επιχειρήσεις μας. Και γι' αυτό πριν αναφέρθηκα και σε ένα πιο ευρύ ρόλο. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό το οποίο μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε πραγματικά ικανοποιητικά μαζί, να κολλάμε μαζί, χωρίς να πλήττεται την εμπιστοσύνη μεταξύ μας, κάθε άλλο. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε την εικόνα του ελέγχου. Και εδώ στο κέντρο μας τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε αναπτύξει αυτό το σύστημα με την τεχνική στήριξη της ΕΜΣΑ που είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια της ναυτιλίας. Είμαστε πρωτοπόροι στον κόσμο γιατί έχει τρία επίπεδα πληροφοριών που προσφέρουμε στα άλλα κέντρα. Η κίνηση των 4.500 ε, σκαφών Βλέπουμε εδώ τη μετακίνησή τους και κάθε μήνα οι πληροφορίες αυτές συγχωνεύονται με το Alert που είναι ο εντοπισμό της θέσης και το IS που αφορά την εμπορική θέση. Έχουμε και αλγόριθμους οι οποίοι μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε πόσο ευάλωτη είναι η κατάσταση όσον αφορά το κάθε σκάφος, πώς δηλαδή επικίνδυνο είναι να δεχτεί επίθεση. Έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας. Κάτι το οποίο μας επιτρέπει να ελέγχουμε και τις τάσεις και να αλλάζουμε την αντιμετώπιση μας ανάλογα με το αν αλλάζουν οι τάσεις. Αν δείτε αυτή τη διαφάνεια θα δείτε εδώ την πορεία των εμπορικών σκαφών βάσει των πληροφοριών που συλλέγουμε. Ποια ήταν το 2013 και ποια το 2015. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τη μετακίνηση των σκαφών στις ακτές της ε, Σομαλίας. Και γιατί, γιατί η απειλή από την πειρατεία έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί η απειλή, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εξακολουθεί να είναι πραγματική. Συνεπώς το έργο μας είναι να συνεργαζόμαστε με την ναυτιλία, με τους εταίρους μας, να παίρνουμε τις πληροφορίες εκείνες οι οποίες μας επιτρέπουν στη συνέχεια να μεταφέρουμε οδηγίες συστάσεις για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μηνύματα λοιπόν. Επόμενη διαφάνεια. Η εξέλιξη του κέντρου ασφάλειας έχει τροποποιηθεί. Βρίσκεται σίγουρα στο κέντρο της επιτυχίας μας. Με το QMTO είναι κεντρικό στην επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι καλύτερες πρακτικές διαχείρισης που εντοπίζονται βοηθούν την ναυτιλία να προστατευτεί και από μόνη της. Και εμείς ως στρατιωτικοί παίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο στις στρατιωτικές συμβουλές που περιλαμβάνονται ε, στο έγγραφο συστάσεων. Πρόκειται για μια αναγνώριση της εταιρικής αυτής σχέσης, γιατί πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και τα τελευταία τέσσερα χρόνια το συντάσσει το κέντρο μας θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Πάντως είναι κάτι που εξακολουθεί να ισχύει και να αποτελεί μια επιτυχία. Εδώ βλέπετε την εικόνα μιας συνάντησης συνεδρίασης SHAPE. Το SHAPE ε, έχει να κάνει με την ε, αποκοινού αναγνώριση κινδύνων λειτουργίες κλπ. 36 τέτοιες συναντήσεις είχαμε τα 6 χρόνια που πέρασαν. Χωρίς καμιά αμφιβολία πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία για το συντονισμό τόσο διαφορετικών στρατιωτικών επιχειρήσεων μαζί. Τρεις φορές το χρόνο συναντιόμαστε στο Μπαχρέιν και εκεί γίνεται ο συντονισμός και η αποκλιμάκωση. Οι συμμετέχοντες στο ΣΕΙΝΤ εξετάζουν το μέγεθός του. Θέλουν να δούνε κάθε φορά πού θα λάβει χώρα το φόρουμ και πώς θα διαμορφωθεί. Η συνεργασία μας με την ναυτιλία όμως όπως σας είπα είναι εξίσου σημαντική. Η ναυτιλία πάντα στέλνει έναν εκπρόσωπο των οργανώσεών της στην συνάντηση αυτή του ΣΕΙΤ. Ακριβώς η συμμετοχή της ναυτιλίας στη στρατιωτική αυτή επιχείρηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όπως ίσως να γνωρίζετε ή να μην γνωρίζετε, Υπάρχει και ένας κλάδος που ονομάζεται περιοχή υψηλού κινδύνου, η οποία έχει μειωθεί αυτή η περιοχή τελευταία. Και στο χάρτη εδώ βλέπετε τα σύνορα της περιοχής αυτής πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα, ότι έχει περιοριστεί δηλαδή αυτός ε, ο χώρος που θεωρείται επικίνδυνος. Μειώθηκε το Δεκέμβριο και αρχίζουμε να έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι αλλάζει η πειρατεία και οι πειρατέ στη συμπεριφορά τους και δεν μας εκπλήσει αυτό γιατί το γεγονός ότι περιορίστηκε ο επικίνδυνος αυτός χώρος σημαίνει για αυτούς ότι η απειλή είναι μικρότερη απέναντί τους. Όπως είπα όμως και πριν, με τα μέσα που έχουμε χρησιμοποιήσει, με την εμπιστοσύνη που έχουμε οικοδομήσει με την αυτιλία, καταφέραμε να πετύχουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε μαζί μας για να διατηρήσουμε την επιτυχία μας. Αυτές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λοιπόν για το μέλλον. Και αυτά είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας όπως σας τα περιέγραψα. Και όλα αυτά μαζί οδηγούν στο να μπορούμε να συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας. Και εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή μου κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θέλω να παρουσιάσω σωστά τον εκπρόσωπο της Επιτροπής είναι ο κύριος Κριστιαν Τιουπάν, ο οποίος είναι αναπληρωτής επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης MOVE στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασχολείται με την αυτιλιακή ασφάλεια. Η... Παρόντες εδώ, αν έχουν μεταξύ τους συζητήσεις, παρακαλώ να το κάνουν χαμηλόφωνα, γιατί μας ενοχλούν. Λοιπόν, κύριε Ντιβάν, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Merci, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρίε και κύριοι. σα ευχαριστώ για την πρόσκληση για να μιλήσω για ένα θέμα καθημερινότητας. Δηλαδή, το πώς θα διασφαλίσουμε τις θαλάσσιες εμπορικές ε, οδούς από την πειρατεία. από την πειρατεία και όχι μόνο. Γιατί η πειρατεία ω όρος χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για ένοπλε επιθέσεις στα πλοία εμπλό. Υπάρχουν όμως βασικές διαφορές έστω και αν στην ουσία μιλάμε για ληστείες Αυτές οι πειρατικές πράξεις είναι αυτές που λαμβάνουν χώρα σε διεθνή ύδατα και οι ένοπλες επιθέσεις συνήθως λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια μιας χώρας. Αυτή η διαφορά λοιπόν είναι σημαντική γιατί αντιμετωπίζουμε τώρα τρεις μεγάλες περιοχές, οι ζώνες όπου αυτές οι πράξεις λαμβάνουν χώρα. ακτές Ομαλίας στα ανοιχτά που σας περιέγραψε ο φίλος Σάμον Τσέρτς γλαφυρά και με, με τρυφροσύνη γιατί αυτά που κάνουν εκεί είναι πολύ επιτυχημένα δυστυχώ. δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού Εκεί λοιπόν έχουμε να κάνουμε με πράξεις πειρατείας που λαμβάνουν χώρα σε διεθνή ύδατα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ένα, ένα ψήφισμα που ανοίγει αυτά τα χωρικά ύδατα στη διεθνή κοινότητα ακριβώς για να παρενέβει και νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα περιθώριο ελιγμού που μας επιτρέπει να καταδιώξουμε τους πειρατές μέχρι τέλους. Μετά έχουμε αυτά που γίνονται στον κόρπο της Γουινέας όπου κυρίως έχουμε ένοπλες επιθέσεις επειδή αυτοί που τις διαπράττουν τον περισσότερο καιρό παραμένουν στο εσωτερικό της επικράτειας των χωρών. Και υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι γι' αυτό. Δηλαδή, το ότι οι χώρες αυτές δεν θέλουν να δουν σκάφη του στόλου, ξένου στόλου για να κυνηγήσουν ακριβώ αυτούς τους ληστέ. Και μετά έχουμε αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Ασία κυρίως με κάποιες υποδιορίσει. Έχουμε τη Σιγκαπούρη και τα στενά του Μάλακα που αποτελούνται κατά 70% από χωρικά ύδατα, από τις γύρω χώρες δηλαδή, όπου έχουμε, όπου έχουμε φαινόμενα κυρίως ένοπλων επιθέσεων, πειρατείας, και μετά έχουμε την ε, θάλασσα της Κίνας, την νότια, όπου έχουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Έχουμε βέβαια πράξεις πειρατείας, ένοπλες επιθέσεις κτλ. Όμως η θάλασσα της Κίνας είναι ουσιώδου σημασία για κάποιε εμπορικέ θαλάσσιε οδού και δέχεται και άλλε απειλέ και άλλες επιβολές αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν με διεκδικήσει εδαφικέ σε σχέση με κάποιε νήσους που είναι εκεί. Εμείς λοιπόν ως Γενική Διεύθυνση Μεταφορών στην Κομισιόν τι εξετάζουμε. Γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τα εμπορικά πλοία αλλά και τα αλλιευτικά που είναι ευθύνη των φίλων μας της Γενικής ΜΑΡΕ. Τα σκάφη μας λοιπόν να μπορούν να πλέψουν, να μεταφέρουν ό,τι πρέπει να μεταφέρουν υπό συνθήκες ασφαλείας κανονικής και κατ' εφαρμογή του θαλασσίου δικαίου που θα πρέπει να είναι αντιληπτό και εφαρμοστό από όλου. δηλαδή η συνθήκη των Ηνωμένων για τη θάλασσα. Πέραν λοιπόν από την Κομισιόν και οι χώρες μέλη και άλλοι οργανισμοί εμπλέκονται για να προσπαθήσουν να πετύχουν κάποια πράγματα και όλοι μαζί συνεργαζόμαστε ώστε να προσπαθήσουμε ανάλογα με την περιοχή να βελτιώσουμε την κατάσταση. Οι παράκτιες χώρες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καταλήξουμε σε αυτό το εντανικό στόχο με πλεύση υποσυνθήκες πλήρους ασφάλειας. Τώρα τεχνικά ή νομοθετικά αν προτιμάτε, τι κάνουμε στην Κομισιόν. Καταρχάς έχουμε έναν κανονισμό σε σχέση με την ασφάλεια των αλληλικών καταστάσεων και των σκαφών που συνδέεται με το ESPS του διεθνού Οργανισμού για τη Θάλασσα Ασφάλεια στις λιμενικέ καταστάσεις και είναι ένας κώδικας ο οποίος λέει ότι όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους και τους φορείς στη θάλασσα, ανάλογα με την σημαία, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση των συνδικών ασφαλείας που θα αντιμετωπίσει το σκάφος κατά τη διάρκεια της πλεύσης ε, του και κατά συνέπεια εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων που θα πρέπει να ισχύουν. Επίσης, από το 2010, 11 Μάρτη, έχουμε μία σύσταση της Κομισιόν που αφορά τα μέτρα αυτοπροστασίας και πρόληψης πράξεων πειρατικών και ενόπλων επιθέσεων κατά των σκαφών. Αυτή η, συνθ... σύσταση καταρχάς ενσωματώνει αυτό που ανέφερε ο Σάμουελ προηγουμένως στα ΜΠΕ και αφορά το σύνολο των καταστάσεων όπου έχουμε έναν κοινό κορμό μέτρων. Ένας από τους στόχους αυτής της σύστασης και της δουλειάς που κάναμε με το BNP και με το, ε, και το MSE, βέλτιστες πρακτικές δηλαδή, και έχουμε καθημερινά πιστοποιητικά συμμόρφωση των ευρωπαϊκών σκαφών θα βρίσκονται σε αυτέ τι περιοχέ. Αυτά τα πιστοποιητικά είναι πολύ σημαντικά γιατί μα επιτρέπουν ακριβώ να διοχετεύσουν αυτέ τι πληροφορίε στι χώρε σημαία, δηλαδή τι ε, αρχέ, τι αρμόδιε των χωρών μελών τη Ένωση και χάρη ακριβώ σε αυτή την φιλική πίεση που ασκούμε στις διοικήσεις το ποσοστό συμμόρφωσης των σκαφών με σημαία χώρου μελών έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά. Γιατί είχαμε πέσει κάποια στιγμή στο 1% ποσοστό που είχε αυξηθεί στο 4-5% αλλά νομίζω ότι εντάξει το ποσοστό είναι αποδεκτό. Τώρα, πέρα από την νομοθετική πτυχή Έχουμε οργανισμούς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ε, Ασφάλεια στη Θάλασσα. Έχουμε να κάνουμε με δεδομένα που αφορούν σκάφη, δεδομένα τα οποία συλλέγονται συνεχώς από την υπηρεσία και τα οποία διατίθενται στους ενδιαφερόμενους. Τι κάνουμε τώρα μέσω μακροπρόθεσμα. Ο τρόπος για να προστατεύσουμε αυτές τις οδούς είναι το να καταστήσουμε αντιληπτό στις παράκτιες χώρες ότι έχουν ευθύνες τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουν και τις βοηθάμε να αναλάβουν αυτές τις ευθύνες. Πώς τις βοηθάμε. Τις βοηθάμε μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης της ικανότητάς τους. Όλα αυτά γίνονται ήδη στο κόλπο της Γουινέας, μέσω της στρατηγικής για το κόλπο της Γουινέας, που υιοθετήθηκε στις 16 Μάρτη του 2015 από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται στη συνέχεια από την Γενική Διεύθυνση Συνεργασίας και Ανάπτυξης και στο κέρας της Αφρικής και στη Σομαλία. Έχω δύο εξέχοντες συναδέλφους στην αίθουσα τον Άρτερ Ιδέα και αποτελεί οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες για τα προγράμματα αυτά από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, επειδή ακριβώς αυτοί τα εφαρμόζουν και οι οποίοι μπορούν να σας δώσουν περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτά από μένα σχετικά με την πρόοδο της κατάστασης. Ξέρω ότι δεν έχουμε περιορίσει το χρόνο, θέλετε λοιπόν θα σταματήσω εδώ και θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω ότι αυτό που έγινε στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας αποτελεί μια θαυμάσια επιτυχία. Δυστυχώς δεν μπορεί να μεταφερθεί αλλού όσο έχει και οι λύσεις για τη Γουινέα και για την Νότια Ανατολική Ασία θα πρέπει να αναζητηθούν με τρόπο διαφορετικό εμείς όμως οπωσδήποτε θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις διαφορετικά η τροφοδοσία μας θα υποφέρει. Ένα στοιχείο. 85% από αυτά που καταναλώνουμε και βρίσκονται γύρω μας κάποια στιγμή έφτασαν φορτωμένα σε ένα πλοίο. Αυτά ένα Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά όπως ανέφερα. Έχουμε και έναν τρίτο ομιλητή, τον κύριο Ζιλ Νόουξ, που δυστυχώς έχασε το τρένο και θα καθυστερήσει. Θα του δώσω το λόγο μετά τον πρώτο γύρο της συζήτησής μας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή. Είχαμε επισκεφτεί το αρχηγείο της επιχείρησης Αταλάντα για να διαπιστώσουμε τη συμβολή της ναυτιλίας στην επιτυχία της συνολικής επιχείρησης. Πολλά θέματα τέθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής μας αυτής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την συγκέντρωση πληροφοριών κατά την συνεργασία ανάμεσα στον τομέα της ναυτιλίας και το αρχηγείο της επιχείρησης Αταλάντα. Γνωρίζουμε ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφάσισαν να χρησιμοποιούν δικά τους μέτρα ασφαλείας στα πλοία. Πώς χειρίζεστε τις ενέργειες αυτές, πώς ε, τις συντονίζετε. Και η τρίτη μου ερώτηση και προς τους δύο μιλητές έχει να κάνει με τα διδάγματα από την επιχείρηση Αταλάντα. και την αξία των εμπειριών. για την ε, επιχείρηση Σοφία. Από ό,τι γνωρίζω, οι παρούσες δραστηριότητες της επιχείρησης Σοφία ε, είναι κυρίως η διάσωση στο πλαίσιο της ε, σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού... του Σόλας, συγγνώμη, ενώ η επιχείρηση Αταλάντα προστατεύει τα συμφέροντα του εμπορικού στόλου. Φαντάζομαι ότι τα εμπορικά πλοία μπορεί να θέλουν να αποφύγουν τις ιδιαίτερα δαπανηρές ε, επιχειρήσεις σόλας. Βέβαια υποχρεούνται σε κάποιο βαθμό με τον ίδιο τρόπο που έχουν υποχρέωση και τα ε, στρατιωτικά σκάφη, αλλά υπάρχουν διαφορές. Τι κοινά σημεία βλέπετε λοιπόν. Ζήτω συγγνώμη, ο κύριος Ντανζόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας και τον κύριο Τυπό που μας υπενθύμησε την τοπολογία του φαινομένου που αντιμετωπίζουμε για την αλήθεια ότι υπάρχει σύγχυση. Στις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Να μην είναι έτσι τυχαία, χωρίς σωστό σχεδιασμό, να μην γίνονται επικαλύψεις. Λοιπόν, για τον κόλπο της Γουινέας, επανέρχομαι σε αυτό. Η εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης ικανοτήτων. Θέλω να μου πείτε, η ΤΕΦΚΟ είπατε κι εσείς ότι το διαχειρίζετε, αλλά έχουμε κάποια τάξη μεγέθους για τον προπολογισμό, για τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται. Τι καλύπτει κατά κάποιο τρόπο ως αρρωγή και προγράμματα για τις ενδιαφερόμενες χώρες. Και κάτι δεύτερο, πιο περίπλοκο ίσως, διπλωματικά τουλάχιστον για να απαντηθεί. Η περίπτωση της Νιγηρίας. Υπάρχει ένα πραγματικό οικονομικό μοντέλο στα ανοιχτά, μακριά από τις ακτές. Υπάρχει εγκληματικότητα στη θάλασσα, οι ομοιρίες. Ξέρουμε ότι από πλευράς ασφάλειας γενικά, αλλά και τις ναυτιλίες πιο συγκεκριμένα, η διάσταση ασφάλειας στην Νιγηρία είναι πάρα πολύ αδύναμη, υπάρχει διαφθορά, είναι περίπλοκο, είναι δύσκολο να δουλεύουμε μαζί τους για την ασφάλεια. Υπάρχει κάποια αξιολόγηση, υπάρχει κάποια πιθανότητα να κάνουμε κάτι αποτελεσματικό μαζί τους για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα στη θάλασσα και η πειρατεία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριος Μπουχνέρ. Σας ευχαριστώ. Μπούχνερ λέγομαι. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία από τις δικές σας ερωτήσεις και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις επιτυχείς επιχειρήσεις, για παράδειγμα της Σομαλίας, των μέτρων που συζητήσαμε εδώ και της προστασίας επί των πλοίων. Από τις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρείες και από τα προγράμματα υποδομής για την καταπολέμηση της φτώχειας των ε, ανθρώπων που ζουν ε, στις ακτές, ε, αφαιρώντας έτσι το πεδίο δράσης των πειρατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη που δεν προέφερα σωστά το όνομά σας, ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ντουπον, έξι πρώην στρατιωτικοί της Βρετανίας κρατούνται, προσπαθούσαν να προστατεύσουν εμπορικά πλοία από πειρατές. Ε, ο Υπουργός Εξωτερικών θεωρεί ότι αυτό είναι ε, αρμοδιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ινδίας, ε, ενώ το διεθνές δίκαιο θεωρεί ότι αυτό είναι θέμα διεθνούς δικαιοδοσίας. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι μόνιμα μέλη, αλλά ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί και πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την κατάσταση των έξι αυτών πρώην στρατιωτικών εάν δώσουμε την αρμοδιότητα του θέματος σε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριο Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόλις αναφερθήκατε στο 85% το ποσοστό. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εμπορικές οδούς και δυναμικό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, η Ινδία, η ε, Νοτιοανατολική Ασία επίσης δραστηριοποιούνται. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον από πολλές πλευρές να υπάρχουν ασφαλείς οδοί. Αναρωτιέμαι αν είναι ρεαλιστικό να έχουμε διεθνή συμφωνία ώστε διάφοροι εταίροι να προστατεύουν, να επιτηρούν, ε, να διασφαλίζουν συγκεκριμένες περιφέρειες και ε, για άλλους ε, ή μαζί με άλλους το κέρας της Αφρικής, στο κέρας της Αφρικής να υπάρχει μόνιμη εποπτεία, περιπολία. να αναθέσουμε στην Ινδονησία ή τη Μαλαισία να προστατεύσουν και τα δικά μας σκάφη και πιο νοτιοανατολικά την Κίνα. Υπάρχουν ε, σχετικοί συλλογισμοί, δηλαδή να γίνει κατανομή των εργασιών για την προστασία διαφόρων περιφερειών και έτσι να μοιράσουμε και το κόστος ε, και ε, την όλη προσπάθεια. Um, ladies mm, Κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Giles Noakes πρώτα. από την BIMCO το Βαλτικό και Διεθνές ε, Θαλάσσιο Συμβούλιο, Συμβούλιο Θαλάσσης και αν υπάρξουν ε, ερωτήσεις θα τις ακούσουμε και μετά θα ε, παρακαλέσουμε και τους τρεις ομιλητές μας να απαντήσουν. Συμφωνείτε? Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νόξ, παρακαλώ. Um, Madam Chair, good morning. ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Στο συγγνώμη που έφτασα αργά. Δεν μπορούσα να φύγω από ό,τι ήθελα λόγω βρετανικών τρένων και γύρω σταρ. Είμαι ο Τζιλ Νόριξ, θα μιλήσω εκ μέρου τη βιομηχανία. Αυτή η παρουσίαση έχει ήδη κυκλοφορήσει στου συναδέλφου στη Ιστορική Τράπεζα όλων των εμπλεκομένων, διεθνέ ε, Θαλάσσιο τάγκ Tank Intercargo, που είναι οι κυριότεροι φορεί εδώ στην εθνική βιομηχανία. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω εδώ, το βρίσκεται εδώ στη διαφάνεια. Θα ήθελα να συζητήσουμε πολύ σύντομα το τι κάνει η βιομηχανία αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσει τις θαλάσσιες οδούς από την πειρατεία πώς αποτρέπεται, αλλά θα μπορούσαμε να ξαναρχίσουμε και φαντάζομαι ήδη έχετε ακούσει κάποια πράγματα και τέλος να υποβάλω μία πρόταση για να αυξήσουμε τη χρήση αυτό που βλέπετε εδώ στη διαφάνεια δηλαδή το ιδιωτικό προσωπικό ένοπλο ασφάλειας και αυτά θα αναφέρω στην διάρκεια της παρουσίασής μου. Επόμενη διαφάνεια. Τι κάνουμε. Προσπαθήσαμε δηλαδή από την αρχή να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες κατευθύνσεις γραμμές για την αποτροπή, αποφυγή και καθυστέρηση της πυρεστίας και περατικών επιθέσεων. Τα τελευταία 8 χρόνια προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και θεωρούμε το κάνουμε επιτυχώς. Έστω και λοιπόν και αν δεν φαίνεται να ισχύει αυτό σε έτη όπως το 2009, 2010, 2011. Σας διαβεβαιώ όμως ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα. Πώς το κάναμε αυτό, μέσω κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών που καθορίζονται σε αυτές τις βελτίες πρακτικές διαχείρισεις που γνωρίζετε εσείς, για τις οποίες είμαστε στην τέταρτη έκδοση τους που παρέχει καθαριτές γραμμές στους πιοκτήτες και στους εμπλεκόμενους στην ασφάλεια για το πώς θα μπορούσαν να διελεύσουν από το Ενδικό Ωκεανό. Περιλαμβάνω επίσης και την ε, συνειδητοποίηση κάποιων στοιχείων ασφάλειας. Είχαμε και μία διάσκεψη που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, όπου συμμετείχαν πολλοί διεθνεί οργανισμοί, ΝΑΤΟ και προσπαθήσαμε λοιπόν να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να γίνει αντιληπτή η απειλή. Μετά, στο κέρας Αφρικής είχαμε ένα κέντρο το οποίο παντρώθηκε από διεθνείς οργανισμούς, βρετανικές υπηρεσίες και το οποίο ενημέρωνε όλα τα σκάφη που περνούσαν από την περιοχή για την κατάσταση που ισχύει εκεί με στρατιωτικέ πληροφορίε όσον αφορά τα σκάφη που περνούσαν από τον ειδικό. Επόμενη διαφάνεια. Τι γίνεται τώρα λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση. Όπω θα γνωρίζετε πολλοί από εσά, η πειρατεία αν πετράπει επιτυχώς σε ένα βαθμό αρκετά επιτυχώς τα τελευταία τρία χρόνια. Και επειδή είναι αδύνατο να κηρύξουμε όλη την περιοχή υψηλού κινδύνου, προσπαθήσαμε να μειώσουμε τον κίνδυνο σε κάποιες περιοχές ε, και αυτό το κάναμε ήδη από το Δεκέμβριο του 2015. Παρ' όλα αυτά θα δείτε ότι ήδη χαρακτηρίζουμε αυτή την περιοχή σχετικά μικρότερη βέβαια αυτή τη φορά, ως περιοχή υψηλού κινδύνου. Περιλαμβάνει τον ε, κόλπο του Αντέν και τη λεκάνη της Σομαλίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αναθεωρούμε όλα αυτά και να τα τροποποιούμε ώστε να αντανακλούν την πραγματικότητα. Αλλά να θυμάστε, η πραγματικότητα αυτή, όπως είπα στην προηγούμενη διαφάνεια, χαρακτηρίζεται από και καθορίζεται τις πληροφορίες που μας παρέχονται και από την ενημέρωση όσον αφορά ε, την πιθανότητα απειλής και την ενημέρωση για την απειλή. Επόμενη διαφάνεια. Ποιε είναι λοιπόν οι πραγματικέ απειλέ όπω ακριβώ αντιμετωπίζονται από τη βιομηχανία σήμερα. Είμαι βέβαιο ότι από την ΑΦΟ, από του Αμοσέρε, θα είχατε κάποια ενημέρωση. Εμεί θεωρούμε συνοπτικά ότι η πειρατεία έχει περιοριστεί αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Η απειλή δεν έχει εξαφανιστεί πλήρω ο κίνδυνος επανεμφάνισης Σομαλών πειρατών είναι υπαρκτός και η παρόνομη αλληλεία στη Σομαλία έχει ανακύψει ως πρόβλημα και αποτελεί ένα σημαντικό καταλήτη για την περαιτέρω επανεμφάνιση της πειρατείας. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι ξέρουμε, η προσπάθεια θα μπορούσε να συνεχίσει να ισχύει, υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν και ευκαιρίες βέβαια, για τους Σομαλούς δηλαδή πειρατές ώστε αυτοί να οδηγηθούν στο να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία. Θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Τι εννοώ. Δυστυχώς, δυστυχώς παραμένει εύκολο τα πλοία αυτά να είναι υπό ομοιρία ιδιαίτερα σε, στις ακτές της Σομαλίας. Αυτό σημαίνει ότι η πειρατεία μπορεί να συνεχιστεί για να υποχωρήσει λοιπόν αυτή η ευκαιρία πειρατείας θα πρέπει να ε, επαγρυπνούμε. Επόμενη διαφάνεια. Πώς ε, καταφέραμε λοιπόν να τα κάνουμε όλα αυτά που πετύχαμε ώστε να μειώσουμε την απειλή και να δημιουργήσουμε μια αποτροπή. Εδώ έχουμε αυτό το τρίποδο που από τρεις πυλώνες. Μπορεί να υπάρχει ένα τέταρτο πυλώνα, το capacity building, αλλά τέλος πάντων δεν διαφωνώ με αυτό αλλά το capacity building, αν αποτελέσει ένα τέταρτο πυλώνα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτούς τους πρώτους τρεις πυλώνες. Πρώτοι τρεις πυλώνες λοιπόν της προσπαθίας μας, οι ναυτικές δυνάμεις, οι βέλτιστες της επαρκής διαχείρισης και η χρήση ιδιωτικού προσωπικού ένοπλου ασφαλείας. Αν αυτά δεν υπάρξουν, τότε δεν υπάρχει συλλογική επιτυχία για την αποτροπή της πειρατείας, όπως λέγαμε, η πειρατεία που υπάρχει ακόμα ως ε, πιθανότητα. Αυτή λοιπόν οι τρεις πυλώνες κατά την απόψη μας είναι απόλυτα απαραίτητη και θα πρέπει να διατηρηθούν προς το παρόν μέχρι να αλλάξει η αξιολόγηση της απειλής. Γιατί η ναυτική παρουσία είναι τόσο σημαντική. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Είμαστε βέβαιοι ότι η αποτροπή ενισχύθηκε από την παρουσία των ναυτικών δυνάμεων. Πριν από αρκετό καιρό, όταν ήμουν στο στρατό, μα είπαν ότι η αποτροπή αποτελείται από ένα μείγμα αξιοπιστία και ορατότητα. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντε. Με την παρουσία λοιπόν ναυτικών σκαφών στην περιοχή υπάρχει ορατότητα, υπάρχει παρουσία που αποτρέπει την πειρατεία σε κάποιο βαθμό. Υπάρχει μια προοπτική λοιπόν ή μια πιθανότητα στρατιωτική απάντηση η οποία αποτρέπει την πειρατεία. Και υπάρχει υψηλό κίνδυνο βεβαίω καταδίωξη των πειρατών, ιδιαίτερα όπω είδαμε το 2010 και 2011. Και μόνο χώρε οι οποίε έχουν επίσημη στρατηγική παρουσία μπορούν να το κάνουν αυτό. Οι ένοπλοι οι οποίοι βρίσκονται στα πλοία δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν έχουν την δικαιοδοσία να το κάνουν. Κάποιο λοιπόν μπορεί να βοηθήσει στην προστασία, αλλά δεν έχει νομική δικαιοδοσία να κάνει κάτι τέτοιο. Οι στρατιώτε έχουν βεβαίω μια συγκεκριμένη δυνατότητα δράση, η οποία αποτρέπει το, την πιθανότητα επιθέσεων στην περιοχή της Αμαλτίας. Η εντολή λοιπόν των στρατιωτικών πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να σταθεί το κατάλληλο μήνυμα προς τους πειρατές και να του αποτρέψει. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Θα ήθελα τώρα να σα πω δύο λόγια για το ένοπλο προσωπικό ασφαλεία στο ιδιωτικό. Γιατί στην βιομηχανία υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία ότι κάποιοι θεωρούν τη χρήση του ω αντικατάσταση ή εναλλακτική λύση τη παρουσία των ναυτικών δυνάμεων. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω το πώς φτάσαμε εδώ. Γιατί δηλαδή τον 21ο αιώνα χρησιμοποιούμε ιδιωτικούς στρατούς ασφαλείας στα σκάφη. Είδαμε ότι χρειάζονται αυτές οι μορφές στρατηγικής παρουσίας ασφαλείας μετά τους πολέμους. Αλλά τώρα βρισκόμαστε σε άλλα όρια, ιδιαίτερα στα ανοιχτή θάλασσα, όπου υπάρχει έλλειψη επιβολή του νόμου και δεν υπάρχει βέβαια μετά από τα χωρικά ύδατα. Οπότε υπάρχει αυτό το φαινόμενο του ασύμετρου πολέμου. Πολύ συχνά υπερτονίζεται από την έλλειψη νομικής υποστήριξης στην ανοιχτή θάλασσα και ο μόνος νόμος είναι το δίκαιο της θάλασσας. Παντού σε όλο τον κόσμο, όχι στον ειδικό ωκεανό μόνο, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό εφαρμογή του νόμου. Δεν είναι ένα κενό που αφορά πόλεμο. Δεν έχουμε να κάνουμε αξιολόγηση με κίνδυνο πόλεμο, αλλά έχουμε να κάνουμε την επιβολή του νόμου. Αν λοιπόν δεν υπάρχει επαρκής αρχική αποτροπή υπό το δίκαιο της θάλασσας, τότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αγοράσουν κατά κάποιο τρόπο ασφάλεια. Είναι μοναδική εναλλακτική λύση όταν αυτές οι πρακτικές διαχείρισεις δεν επαρκούν. Και όπως οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, όταν πρέπει να αγοράσετε κάτι, κάνετε κάποιες ρυθμίσεις εμπορικές. Αυτές οι εμπορικές ρυθμίσεις μετά ενισχύθηκαν παραδόξως από ένα συμβόλαιο από μια σύμβαση των Guardcom για να προστατευτεί και το πλήρωμα αλλά και ο πλειοκτήτης από αυτούς τους κινδύνους. Υπάρχει όμως ένας άλλος κίνδυνος το να θεσμοποιηθεί αυτό, αυτή η σύμβαση για διάφορους λόγους. Επόμενη διαφάνεια. Κίνδυνο ανάλυση. Συγγνώμη. Ανάλυση κινδύνου. Τελευταία λύση. Θα πρέπει οτιδήποτε κάνουμε εδώ να διέπεται από την ανάλυση του κινδύνου. Ο κύριος παράγοντα εδώ είναι ο νόμος και το χρησιμοποιώ αυτό για να εξηγήσω ότι ένα σκάφος το οποίο έχει χαμηλή ταχύτητα, κάπου, κάτω από 18 κόμβους ή 10 κόμβους. Είναι πολύ ευάλωτος στόχος, ανεξάρτητα από όσους, από όσους βάλετε ένοπλους στο πλοίο ή χρησιμοποιείτε αντιλίες ή οτιδήποτε άλλο έξιμο το οποίο έχει αναπτυχθεί για την προστασία από τους πειρατές. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν το λόγο οι ένοπλοι φύλακες εντάσσονται εδώ σε αυτή την ανάλυση κινδύνου που, την οποία θα πρέπει να κάνει ο πλειοκτήτης. Ένα παράδειγμα σήμερα αυτού του φαινομένου και τη συνεχή χρήση του, τους ε, είναι το ότι 80% των σκαφών που περνάνε από τη λεκάνη τη Ομαλία, χρησιμοποιούν ένοπλου φυλακέ, γύρω όμω το 20% πέρα τη ζώνη των 65 μοιρών ανατολικά. Γιατί εδώ ακριβώς εξαρτώμαστε από την ανάλυση κινδύνου. Όσο πιο κοντά πάμε στη λεκάνη της Ομαλία, πιο ψηλός ο κίνδυνος. Αλλά αν θέλουμε ω διεθνή κοινότητα να συνεχιστεί το εμπόριο σε αυτό το κομμάτι της Αφρικής, αυτό θα πρέπει να, να κάνουμε, να ανοίξει το Μαγκαντήσου και άλλα λιμάνια στην Σομαλία για να βελτιώσουμε το εμπόριο με την Τανζανία και την Κένια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε από τη λεκάνη Σομαλία. Σομαλίας. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Εμεί λοιπόν θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση των ενόπλων φρουρών και δεν αποτελούν μια χρήση λύση γιατί στην ουσία μειώνουμε την πραγματική αποτροπή δεν υπάρχει δυνατότητα δίωξη η άσκηση δίωξης στους πειρατές και μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε έλλειψη, έλλειψη μάλλον οποιαδήποτε στιγμή ένοπλων φυλάκων. Γιατί αν φύγει η ναυτική παρουσία, η στρατηγική παρουσία, το θα αλλάξει βέβαια και η αναξύλωση κινδύνου των πλειοκτητών. Ίσως μπορεί να υπάρξει βεβαίως και μια μεγάλη αύξηση αυτών, του, αυτών των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν θα ήταν και πολύ θετικό. Ίσως τα θέματα αυτά θα έπρεπε να συζητηθούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Θάλασσα, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση σε σχέση με την ύπαρξη αυτών των πλωτών ένοπλων ομάδων. Και δεν ξέρω κατά πόσο κάποιοι θεωρούν ότι αυτό πρέπει να κατασταθούν και στου λιμένε, αλλά βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό να αυξάνεται. Υπάρχουν βεβαίω και ζητήματα νομικά και οι διακλαδώσει του, όπω α πούμε οι κανόνε για τη χρήση βία από ένα ενόπλο φρουρό. Υπάρχουν διάφορε ε, μορφέ αυτή τη παρουσία και αυτού του φαινομένου που αφορά, α πούμε, το δίκαιο τη θάλασσα και τη σημαία ευκαιρία. Υπάρχουν νόμοι, αλλά βεβαίω ποικίλουν πολύ σημαντικά και αυτό σήμερα συνεχίζει να αποτελεί ένα πρόβλημα όσον αφορά τους πλειοκτήτες. και αυτό αποτέλεσε και ένα από τους κύριους λόγους της σύναψης αυτής της σύμβασης GATCOM. Και υπάρχει βέβαια και ένα σοβαρός λόγος ανησυχίας για την κλιμάκωση της βίας. Αν ξαφνικά ε, φύγει η στρατιωτική παρουσία και αν δούμε ότι υπάρχουν κινήσεις επιθετικές ε, προς τα πλοία, και αυτό το βλέπουμε τους τελευταίους μήνες συνεχώς, αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς βία για να αποτρέψει τη βία, τότε μπορεί κανείς να καταλήξει μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Ιδιαίτερα αν θα πρέπει να λάβει υπόψη του κανείς και τους ε, ε, τίγρες τα Μίλ, που συνήθως πυροβολούνται ή καταδιώκονται από τα κυβερνητικά σκάφη όταν καταλαμβάνουν αληφτικά σκάφη. Και αυτό είναι ως κατάσταση πολύ επικίνδυνο και δεν θα θέλαμε να το δούμε. Δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα ασφάλειας και ίσως να υπάρχουν εδώ και ιστορικοί λόγοι που ευχαριστώ να συζητήσω αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Υπάρχουν εδώ κάποια κύρια μηνύματα που θα ήθελε να στείλει η βιομηχανία στην Επιτροπή σας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επίσημη προσπάθεια, ανυποχώρητη και αποτελεσματική. Όσον αφορά τώρα τις εντολές, μια σοβαρή διεθνής παρουσία με λογοδοσία θα πρέπει να διασφαλίσει ακριβώς την αποτροπή της επιστροφής των πειρατών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και άλλα μέτρα να, ώστε να προστατεύσουμε τα σκάφη μετά από μια διεξοδική ανάλυση κινδύνου. Θα υπάρξουν αλλαγές βέβαια σαν αφορά τη διεθνή παρουσία, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για αυταρέσκεια από όλου τους εμπλεκόμενους και του ενδιαφερόμενους σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Αυτά προηγουμένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας, ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τους προσκεκλημένους μας σχετικά με την κατάσταση στην Δυτική Αφρική. Ναι, πράγματι έχει μειωθεί η πειρατεία στο κέρας της Αφρικής, ιδιαίτερα από την Σομαλία. Βλέπουμε όμως αύξηση της πειρατείας στην Δυτική Αφρική και πολλά πλοία στα οποία έχουν γίνει επιθέσεις από πειρατές όχι μόνο στην Ιγυρία που κατά κάποιο τρόπο είναι παλιά ιστορία μιλάω όμως για την ακτή Ελεφαντοστού, την Γκάνα, την ε, Γουινέα, το Τόγκο και το Μπενίν. Οι πειρατές αυτοί δεν καταλαμβάνουν τα ε, πλοία και ζητάνε λίτρα μετά αλλά κλέβουν τα αγαθά, πετρέλαιο κλπ πώς αντιδρά η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα αυτή πρόκληση, η οποία γίνεται όχι μόνο απειλή, αλλά θέτει και διάφορα οικονομικά θέματα. Αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν διπλασιάσει τα ασφάλιστρα για τα πλοία που ταξιδεύουν στη Δυτική Αφρική. Όλα γίνονται πιο ακριβά. Αυτή είναι σημαντική απειλή και για τις οικονομικές συναλλαγές μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα και στους τρεις ομιλητές μας να απαντήσουν στις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Δυστυχώς κύριε Νόξ δεν ακούσατε τις ερωτήσεις που τέθηκαν νωρίτερα. Ε, εάν ε, θελήσετε να πάρετε το λόγο αργότερα θα σας παρακαλέσω θα παρακαλούσα τον ε, κύριο Σόμος να πάρει το λόγο πρώτος, μετά ο κύριος Εντυπών και ο κύριος Νόξ. Ε, δυστυχώς θα πρέπει να αφήσω το βήμα ε, για πέντε λεπτά. Ε, την Προεδρία στον κύριο Γκάλερ. Ε, σας ευχαριστώ. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις κατά την πρώτη κατά τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και ίσως μπορούν οι συνάδελφοί μου να με βοηθήσουν ιδιαίτερα όσον αφορά την Δυτική Αφρική που δεν, είναι, δεν ανήκει στον τομέα εμπειρογνωμοσύνης μου. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την πρώτη ερώτηση όσον αφορά την ανταλλαγή ε, μυστικών πληροφοριών. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που προέρχεται από τον τομέα της ναυτιλίας, διότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μία από τις βασικές επιτυχίες μας ε, όσον αφορά την καταστολή της πειρατείας ήταν οι πληροφορίες που λαμβάναμε από καπετάνιο του πλοίου την ώρα της πειρατείας. Έτσι λοιπόν οι ε, ναυτικές δυνάμεις μπορούσαν να αντιδράσουν γρήγορα και αυτό ήταν θεμελιώδης παράγοντας. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις ε, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης, τα BMP, ε, ως σημείο αναφοράς. Δηλαδή τα σκάφη θα πρέπει προαιρετικά να μας δίνουν όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες την στιγμή που βλέπουν ε, να υπάρχει κάποια απειλή, διότι μιλάμε για τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις. Δεν είναι mm. τόσο σημαντικό το θέμα αυτό τόσο πια. Συνεχίζει όμως να αποτελεί σημαντικό μέρος ε, της ανταλλαγής πληροφοριών μας με τον ναυτιλιακό τομέα. Επίσης όσον αφορά τα διδάγματα από διάφορα μέρη του κόσμου ε, σε σχέση με την επιχείρηση Σοφία στην Μεσόγειο. Ακούστηκαν και λεπτομέρειες σχετικά με την EUNAFOR και την επιχείρηση Σοφία και την επιχείρηση Αταλάντα. Είναι αρκετά διαφορετικές οι λεπτομέρειες. Ε, θα επιτρέψω στους συναδέλφους να σχολιάσουν τις επιχειρήσεις αυτές. Θα πρέπει όμως να τις αντιμετωπίσουμε διαφορετικά, διότι ε, αυτό που κάναμε στον Ινδικό ωκεανό βασίστηκε στην εμπιστοσύνη. Με άλλα λόγια, ε, λαμβάνουμε πληροφορίες από έναν καπετάνιο για να προστατευτεί από μια απειλή. Και εξαρτάται λοιπόν, περιμένει μια αντίδραση. Γι' αυτό μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό αποτελεσματικό στον Ειδικό ωκεανό. Στην Μεσόγειο όμως το συμφέρον του, καπετάνιου δεν έχει να κάνει με ε, την προστασία του σκάφους, το έχει να κάνει με μια υποχρέωση την, ε, ε, την οποία πρέπει να εκπληρώσει. Είναι λοιπόν σημαντικό να βρούμε έναν τρόπο ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Μία ερώτηση στην οποία επίσης θα ήθελα να απαντήσω. Ακούστηκε και είχε να κάνει με τις διεθνείς συμφωνίες για την εποπτεία. Ε, ακούστηκε η δυνατότητα συνεννόησης με την ε, Κίνα ε, ή την ε, Ινδονησία. Θα ήθελα να πω ότι συνεργαζόμαστε με αυτές τις χώρες, ε, με ε, τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για να βελτιώσουμε την εποπτεία. Θα ήθελα λοιπόν απλά να πω για τα πρακτικά ότι πράγματι υπάρχει τέτοια συνεργασία στρατιωτική. Θα ήθελα να κλείσω εδώ και να δώσω την ευκαιρία στους συναδέλφους να απαντήσουν σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο Ντυπών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε στους pickups που είναι οι ιδιωτικοί φύλακες στα σκάφη. Ε, ήταν κάτι που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς και ήταν μια απάντηση τι μάθαμε όμως, ποια ήταν τα δάγματα από την Αταλάντα ρωτήσατε. Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Σάιμον. Εμείς μάθαμε ότι χωρίς εμπιστοσύνη ανάμεσα στους εφοπλιστές και τις αρχές, τους πλειοκτήτες και, τους, και τις αρχές, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν όλοι ότι οι πληροφορίες τους, τα δεδομένα τους δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για μια στρατιωτική αποστολή υπέρ της προστασίας τους. Αν δεν έχουν αυτή τη διασφάλιση δεν γίνεται τίποτα. Το δεύτερο δίδαγμα που πήραμε ήταν ότι με καλή θέληση, και εδώ απαντάω και στον κύριο Γκάλερ, με καλή θέληση λοιπόν μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιο είδους αμοιβεοποίηση. οπορτινουστική που θα μπορούσατε να πείτε, ευκαιριακή, υπέρ των χωρών εκείνων που έχουν συμφέροντα στην περιοχή και θέλουν να πάνε όλα καλά στην περιοχή. Και θα έλεγα μάλιστα ότι ακριβώς και αυτό είναι και το όριο της λεγόμενης αμοιβοποίησης. Ο ένας βοηθά τον άλλον. Και απαντάω στον κύριο Γκάλερ ότι αν δείτε τι γίνεται στην Νοτιοανατολική Ασία, διαπιστώνετε ότι δύο κύριοι παράγοντες στην περιοχή, η Ινδονησία δηλαδή και η Μαλαισία, δεν είναι μέλη της περιφερειακής δομής RICAP, όπως ονομάζεται. Και αυτή η δομή έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το φαινόμενο, που λαμβάνει η χώρα μπροστά στα μάτια τους. Και όμως αρνούνται να συμμετέχουν σε αυτήν τη δομή, ενώ στη ρίκα συμμετέχουν περίπου όλες οι χώρες από την Ινδία μέχρι την Νότια Κορέα. Υπάρχουν λόγοι υπερβολικού εθνικισμού από ό,τι φαίνεται που έχουν σαν αποτέλεσμα οι δύο αυτές χώρες να μην θέλουν να συμμετέχουν. Δεν είναι κανένα μυστικό, είναι γνωστό ότι σπάσει ότι οι δύο αυτές χώρες είναι ανάδελφες. Και ακριβώς εκεί είναι που συμβαίνει και το πρόβλημα. Στρέφομαι τώρα προς τον κύριο Ντανζό. Το θέμα του προϋπολογισμού, τι θα διαθέσει ντεύκο δηλαδή για τον κόλπο αυτό. Ο συνάδελφος που είναι εδώ στην αίθουσα μπορεί να σας απαντήσει πολύ καλύτερα από μένα, οπότε ο πρόεδρος αν θέλει μπορεί να του δώσει τον λόγο μετά. Όσον αφορά πάντως την κατάσταση στην Ιγυρία, δύσκολα μπορώ να επεκταθώ. Όμως θα σας ε, κάνω μία μεταφορά. Αν ο νευτιλιακός κλάδος νιώσει ότι πρέπει ο ίδιος να δημιουργήσει ένα κέντρο ε, κατανομής των πληροφοριών, το ΕΝΤΙΣ, ξέρετε ότι για κάθε πλειοκτήτη ένα ευρώ είναι ένα ευρώ, δεν πρόκειται να δαπανίσει αν ε, δεν είναι αναγκαίο αν δεν έχει κάποιο συμφέρον να το κάνει. Αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχει πρόβλημα με την διανομή της πληροφορίας και με το συντονισμό στην περιοχή. Και για να είμαι εντελώ ξεκάθαρος μαζί σας, συζητήστε με όποιον πλειοκτήτη θέλετε, μικρό ή μεγάλο. Όλοι θα σας πούν, οι πιο ευγενείς τουλάχιστον, ότι έχουμε πολλές δυσκολίες να δίνουμε πληροφορίες στις χώρες που έχουν ακτές, όταν έχουμε βρεθεί σε δύσκολη θέση. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Για να επανέλθω τώρα στη Μεσόγειο και σε αυτό που ρωτήσατε εσείς κυρία Πρόεδρε για τη συμπεριφορά των εμπορικών πλοίων όταν προχωρούν σε επιχειρήσεις διάσωσης ναυαγών. Για ένα πράγμα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον εμπορικό στόλο. Και αυτό είναι το ότι δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του. Είτε πρόκειται για τη σύμβαση όλες είτε πρόκειται για την ηθική υποχρέωση που έχει. Και ειλικρινά υπήρξε δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα με διορθώσει και ο Giles. Δεν ξέρω ποιος ήταν εσύ, την έκανε αυτή τη δήλωση κάποιος άλλος που έλεγε ότι ο νευτιλιακός ο κλάδος δεν χρειάζεται να του το πει κανείς για να αναλάβει τις ευθύνες του όταν πρόκειται για τη διάσωση ναυαγών γιατί είχε αναφερθεί ότι ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει αντισταθμίσματα κτλ. Οι πλειοκτήτες ήταν ξεκάθαροι και είχαν πει όχι, είναι δικιά μας ευθύνη. Αν δεν σεβαστούμε αυτό, τότε δεν σεβόμαστε πια τίποτα. Αλλά ο Τζάιλς θα μπορέσει ίσως να πει περισσότερα γι' αυτό. Η πρόεδρος. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε να παρέμβω εδώ, λέει πρόεδρος. Συγγνώμη. Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι η επιχείρηση γίνεται ως επιχείρηση σόλας τώρα. Και μπορώ να φανταστώ ότι όταν πρόκειται για κάτι μαζικό και συνεχιζόμενο φαινόμενο, τότε μπορεί αυτού του είδους οι περιοχές, η λεκάνη της δηλαδή, να αποφεύγεται από τα εμπορικά σκάφη. Δεν είπα ότι η εμπορική ναυτιλία εγκαταλείπει επιχειρήσεις όλας. Έτσι, ήθελα να το διορθώσω αυτό για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ευχαριστώ. Όντως έτσι σας είχα καταλάβει, πράγματι. Αλλά για να σας απαντήσω τότε εντελώς ρεαλιστικά. Αυτοί που έχουν μια θαλάσσια διαδρομή που περνάει από την κεντρική Μεσόγειο, το κάνουν για εμπορικούς <coughs> λόγους. Και θα συνεχίσουν. Γιατί αν δεν περνούν από την κεντρική Μεσόγειο, αυτό σημαίνει ότι δεν περνάνε από τη διόρυγα του Σουές, αυτό σημαίνει ότι κάνουν το γύρο της Αφρικής τρεις μέρες παραπάνω δηλαδή στη θάλασσα με όλο το επιπλέον κόστος που σημαίνει αυτό. Οπότε όχι. Σίγουρα Τζάιλ θα μιλήσεις και εσύ γι' αυτό. Για τον κόλπο της Γουινέας τώρα και την ερώτηση σχετικά με αυτό του κ. Τζοφρέτα. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, υπάρχει μια στρατηγική, υπάρχει διπλωματική κινητικότητα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών, προκειμένου οι χώρες που είναι εκεί στις ακτές να αναλάβουν τις ευθύνε τους. Τις στηρίζουμε με διαδικασίες βέβαια μακρόχρονες και περίπλοκες. Η περιοχή αποφάσισε να έχει μια διάσκεψη των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων που θα έπρεπε να λάβει χώρα στην πόλη Λομέ στις 15 Οκτωβρίου που μας έρχεται. Και θα είναι αφιερωμένη η συνάντηση αυτή σε αυτό το θέμα. Είχε προγραμματιστεί ήδη για πέρυσι, αλλά ήταν τόσο περίπλοκο για τους Αφρικανούς φίλους να οργανώσουν την εκδήλωση αυτή που δεν έγινε. Παρά λοιπόν την βοήθεια που τους προσφέρουμε, δεν θα έλεγα ότι βλέπουν διαφορετικά τον παράγοντα χρόνο εκεί, αλλά αντιμετωπίζουν διαφορετικές προτεραιότητες. Έτσι δεν βλέπουν απαραίτητα την κατάσταση όσον αφορά την ε, προστασία ε, στη θάλασσα με τον ίδιο τρόπο ε, που τη βλέπουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Με δύο λόγια, αν έχουν να διαλέξουν, να χτίσουν ένα σχολείο, ένα δρόμο ή να χρησιμοποιήσουν ναυτιλιακά μέσα για να αντιμετωπίσουν ενδεχομένω τους πειρατές, η επιλογή που θα κάνουν θα είναι πάρα πολύ εύκολη, θα χτίσουν το σχολείο, θα φτιάξουν το δρόμο. Και επιβεβαιώθηκε αυτό και σε ένα σεμινάριο που βρεθήκαμε και οι μας, όπου ο κύριος σύμβουλος ε, του Προέδρου της Δημοκρατίας ε, της Εκτής του Ελεφαντοστού το κατέθεσε πολύ συγκεκριμένα. Ωραία, νομίζω ότι μίλησα για όλα τα ζητήματα, αλλά να επανέλθω στην ερώτηση του κύριου Μπουχνέρ για την διάρθρωση των μέτρων αυτοπροστασίας pickups και ναυτιλιακές ε, επιχειρήσεις. Πρέπει να επανέλθω στο παράδειγμα που έδωσε ο Τζάιλς για αυτό το σκαμνί με τα τρία πόδια που αν λείψει το ένα, το σκαμνί δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Προτού να δώσω το λόγο στον κύριο Νόξ, να του θέσω τη δική μου ερώτηση. Να την κάνω πιο σαφή μάλλον. Μάλλον θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό και ε, σε διαφορετικό σχηματισμό. Στην ε, προηγούμενη συνάντησή μας ο κυβερνητής Σμιθ μας παρουσίασε την επιχείρηση Αταλάντα. παρακολουθούμε από κοντά την ε, επιχείρηση αυτή και εκτιμούμε ιδιαίτερα τα επιτεύγματα της επιχείρησης αυτής. Η εμπειρία της Αταλάντα μας κάνει να θέλουμε να διευρύνουμε ε, το πεδίο εφαρμογής της αποστολής ε, EUNAFOR. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιχειρήσεις σόλας. Στο μέλλον θα θέλαμε να μπορούμε να σταματήσουμε την ε, λαθρέα διακίνηση ανθρώπων η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι διδάγματα μπορούμε να εξάγουμε και εγώ τυχαία προέρχομαι από τον τομέα της ναυτιλίας Οπότε είμαι η τελευταία που θέλω να προσβάλλω τον τομέα αυτό. Νομίζω ότι υπήρξε παρανόηση αλλά σίγουρα είναι δύσκολο για μας να συγκρίνουμε μεταξύ τους ε, τις δύο αυτές επιχειρήσεις, διότι η ουσία των δύο αυτών επιχειρήσεων είναι πολύ διαφορετική. Προσπαθώ να αξιολογήσω λοιπόν ε, την συμβολή του τομέα της ναυτιλίας και στις επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Παρεπιπτόντος, ο κύριος Σμιθ ε, μας είπε ότι πρόσφατα ε, πραγματοποιούνται και περισσότερες προσπάθειες από πλευρά της Σόλας ε, στον κόλπο του Άντεν λόγω της Γεμένης και της μετανάστευσης εκεί. Αυτό λοιπόν περιπλέκει όλο το θέμα. Σας δίνω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ζητώ συγγνώμη αν δεν σας ε, αποκάλεσα με τη σωστή ονομασία. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας ε, και καταλαβαίνω και τι εννοούσε ο συνάδελφος ο κύριος Σοντιπών, τον οποίο γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει η απέτηση ένα εμπορικό πλοίο να βοηθήσει οποιοδήποτε άλλο σκάφος αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ε, ο καπετάνιος θα το κάνει αυτό διότι μπορεί να βρεθεί ο ίδιο στη δύσκολη θέση κάποια άλλη μέρα. Ε, ωστόσο, στη Μεσόγειο υπάρχουν σημαντικά προβλήματα διότι όταν εκπονήθηκε η Συμφωνία Σόλας δεν εκπονήθηκε στο πλαίσιο ε, μικτής μαζικής μετανάστευσης και έτσι λοιπόν τώρα ο τομέας της ναυτιλίας αντιμετωπίζει προβλήματα διότι δεν περίμενε ποτέ να πρέπει ε, να συμμετέχει τόσο πολύ στο θέμα αυτό. Ε, κυρία Πρόεδρε και ο κύριος Σεντυπών θα σας πει ότι πάντα ε, αντιδρούσαμε όπου έπρεπε και επίσης συχνά μας έχουν ζητήσει να πάμε σε κάποιο κέντρο, ε, ε, σε κάποιο αρχηγείο και τελικά δεν μας χρησιμοποίησαν. Ε, Παρ' όλα αυτά ευχαρίστως θα το κάνουμε αυτό, διότι... Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του προγράμματος διάσωσης, διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος του τομέα ναυτιλίας και μάλιστα καταβάλλονται πολύ μεγάλες προσπάθειες σε όλες οι ε, παρούσες επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιούνται εδώ και δύο χρόνια έχουν ε, μειώσει, δεν θυμάμαι τον αριθμό της συγκεκριμένη επιχείρησης, συγχωρήστε με, αλλά με την ε, αντικατάσταση του επιχειρησιακού προγράμματος που υπήρχε ε, πριν ε, δύο χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των εμπορικών σκαφών από τα οποία ζητήθηκε βοήθεια. Επίσης γίνονται προσπάθειες για να μειωθεί η λαθρέα διακίνηση και ακριβώς γι' αυτό λιγότερα πλοία χρειάστηκε να αποκλίνουν από την πορεία τους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο τομέας της ναυτιλίας είναι πιο διατεθειμένος να βοηθήσει. Μας ρωτήσατε τι διδάγματα ε, μπορούμε να εξάγουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Η πιο σημαντική είναι ε, η επικοινωνία και ο συντονισμός. Όπως εξήγησαν οι συνάδελφοί μου, ε, το πρόβλημα είναι τελείως διαφορετικό τώρα και γι' αυτό πολλά από τα διδάγματα αυτά δεν μας βοηθάνε πια. Έχουμε όμως ε, αυτήν την εξαιρετική ε, σχέση με την ε, MSCHOA και να επαναλάβω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιχείρηση Αταλάντα αλλά η σχέση αυτή δεν υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτός είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους που καταφέραμε να προχωρήσουμε και να αποτρέψουμε την πειρατεία σε μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα και κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συμμετέχουμε εξίσου ανοιχτά. Έχουμε ε, επαφές με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και με το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την επιχείρηση Σοφία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων πραγματοποιείται στην Ιταλία και με την Κονφιτάμα, το εμπορικό ναυτικό επιμελητήριο. Θα ήθελα όμως να καλέσω την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλέσει τον διεθνή τομέα της αλίας να συμμετάσχει πιο ενεργά για να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και να μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα όταν αντιμετωπίζουμε καταστροφή. Έχει εκπονηθεί ένα φυλάδιο προς τους καπετάνιους ε, σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σύμφωνα με την Σόλας. Είναι αρκετά ογκώδες ε, το υλικό αυτό και νομίζω ότι θα είναι δύσκολο ε, να ε, το διαβάσει ο καπετάνιος σε περίπτωση κρίσης. Εμείς έχουμε φτιάξει μία κάρτα που μπορεί να έχει ο καπετάνιος στη γέφυρα που δίνει απλές οδηγίες σε περίπτωση προβλήματος. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια απειλή, πρέπει να τη γνωρίζουμε, είναι παγκόσμια η απειλή αυτή και παρακολουθούμε στενά την ε, απειλή της τρομοκρατίας και φοβούμαστε διότι ένα κράτος ε, σημαίας έχει ζητήσει από τα σκάφη του να αυξήσουν κατά πολύ τα μέτρα ασφαλείας σε ένα μέρος της Μεσογείου. Αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και είναι έλλειψη ε, κατανόησης, είναι παρερμηνία του κώδικα ISPS, διότι εάν λάβει κανείς κάποια κλίση ε, να βοηθήσει σε διάσωση και πρέπει να αποκλίνει από την πορεία του, ε, τι θα πρέπει να κάνει, διότι ε, αντιμετωπίζει δύο καταστάσεις αντιφετικές σε σχέση με τη συνθήκη Σόλας. Γι' αυτό ακριβώς ο ναυτιλιακός τομέας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επιχείρηση Σοφία και πολύ ευχαρίστω ε, θα συμμετάσχουμε. Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω αυτό να απαντάει τη δική σα και άλλε ερωτήσει ε, για την ε, Μεσόγειο. Έχω και κάποιε άλλε παρατηρήσει, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Νομίζω ότι ε, έπιασα, το, έπιασα ζουμί των περισσότερων ερωτήσεων. Οι τελευταία στην οποία αναφέρθηκε ο Κρίστιαν, νομίζω ότι απάντησα πολύ καλά, αλλά ευρωβουλευτής ακόμα έχει ε, αμφιβολίες ε, μπορεί να ε, κοιτάξει τις διαφάνειές μου αλλά είναι τελείως παράλογο η διεθνής κοινότητα να ζητάει από τον αυτιλιακό τομέα να διασφαλίσει τη δική του ασφάλεια διότι πιθανότατα να υπάρχει σύγκρουση δικαιοδοσιών και κάποια κράτη-μέλη να περιθωριοποιηθούν και να βρεθούν υπό ισχυρή πίεση αν συμβεί κάτι τέτοιο. Φοβάμαι ότι η κλιμάκωση θα είχε σημαντικές συνέπειες και για την καθετερία και για το προσωπικό του πλοίου. Ε, αντιμετωπίζουμε λοιπόν δύσκολες καταστάσεις. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα πλοία και ε, προσωπικά τους, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς ε, μέσα στην αίθουσα αυτή δεν βλέπει ε, το μέλλον της ε, ναυτιλίας με ένοπλους φρουρούς στα εμπορικά σκάφη. Έτσι πάμε πίσω στο παρελθόν. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, συμφωνώ πολύ με τον συνάδελφο. Νομίζω ότι απαντήθηκε πλήρω η ερώτηση αυτή. Και το μόνο άλλο θέμα που τέθηκε και καταλαβαίνω ότι μιλάτε για όλες τις θαλάσσιες οδούς, η Δυτική Αφρική αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με την Σομαλία, όπως δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με την Νότιο-Ανατολική Ασία. Κάθε περιοχή έχει δικά της, δικές της ιδιαιτερότητες και δικά της προβλήματα. Ωστόσο, όπως είπε ο κύριος Ντυπον, ε, το γεγονός είναι ότι έχουμε αναγνωρισμένα κράτη των Ηνωμένων Εθνών με δική τους νομοθεσία, δικά τους ε, εδαφικά ύδατα και δικές τους οικονομικές ζώνες και γι' αυτό θα πρέπει να τα σεβαστεί ο τομέας της ναυτιλίας. Δεν μπορεί να ε, παραβιάζει αυτούς ε, τους νόμους και ακριβώς γι' αυτό δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα διδάγματά μας από την Σομαλία σε άλλα μέρη. Ακόμα και η χρήση μη οπλισμένων φρουρών σε νιγηριανά ύδατα δεν γίνεται καλά αποδεκτή και ε, η Νιγηρία πρέπει να πληρώσει κανείς για την δική του προστασία ε, σε εδαφικά ε, ύδατα κάτι που δεν συνάδει με την συνθήκη UNCLOS και κατά την ταπεινή μου γνώμη η συνάντηση που, πραγματοποιήθηκε, που ε, προγραμματίστηκε για το Τόγκο όπου πιστεύω ότι θα παρευρεθούν υπουργοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει οι παράγοντες που θέλουν να λύσουν το θέμα αυτό και αυτό δεν ε, συμπεριλαμβάνει μόνο ε, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη του κόλπου της Γουινέας και θα πρέπει να υποχρεώσουμε τα κράτη αυτά να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη συνθήκη UNCLOS διότι εάν το κάνουν αυτό, τότε λογικά θα είναι αδύνατον να συνεχιστεί η πειρατεία. Αλλά, όπως έχω πει επανειλημμένα, εάν υπάρχει ανομία ε, στη στεριά θα υπάρχει και στη θάλασσα. Και γι' αυτό εναπόκειται σε φορέα πιο μεγάλο και πιο ισχυρό από τον τομέα της ναυτιλίας να κάνει τα δέοντα, να πράξει τα δέοντα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει σε υπερεθνικό επίπεδο, για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένα Έθνη με ψηφίσματα του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν απαντά στην ερώτησή σας, αλλά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο, αλλά κατάλαβα ότι δεν απάντησα στο ερώτημα του κ. Κέν σε σχέση με τους έξι Βρετανούς υπηκόους που είναι φυλακισμένοι στην Ινδία. κ. ρώτησε τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν. Δυστυχώς δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη μας για αυτό το συμβάν όπως κάναμε και κάνουμε για τους δύο ναύτες του Ιταλικού ναυτικού που βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση στην Ινδία. Δυστυχώς το θέμα αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε μια νέα υπηρεσία, την εξωτερική υπηρεσία εξωτερικής δράσης, που έχει αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι σε συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη χώρα, την Αγγλία και την Ιταλία, θα κάνει κάτι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. για να μην ε, εμποδίζει η του ενός της πράξης του άλλου. Και οι Ινδικές αρχές είναι έτσι πολύ ευαίσθητες σε θέματα εθνικής κυριαρχίας. Αυτά πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις παρουσιάσεις. Νομίζω ότι μας ικανοποίησαν οι απαντήσεις. Δεν υπάρχει άλλος γύρος ερωταπαντήσεων, οπότε να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τους συγγητές μας, παρά τα προβλήματα τα σιδηροδρομικά, καταφέραμε να συζητήσουμε το ζήτημα σε βάθος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. τώρα θα έχουμε στη συνέχεια μια σημαντική ακρόση για την ΑΦΕΤ. Αυτά από εμά. Ευχαριστώ. Γεια σας.